Ας ξεκινήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ρέτζι και πάμε στην υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης. Ένα σύντομο σχόλιο έχω να κάνω εγώ για την ημερήσια διάταξή μας. Συγχαίρω την κυρία Κρέτσου. Είναι και πάλι εδώ μαζί μας για να ανταλλάξουμε απόψεις με τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζη, αλλά θα πρέπει να φύγει στις 4 και 4. Σωστά? Επειδή υπάρχει έκτακτη συνεδρίαση του Κολεγίου των Επιτρόπων. Οπότε, με αυτή τη μικρή αλλαγή, μπορούμε να συνεχίσουμε την συνεδρίασή μας. Δώστε μας παρακαλώ κύριε Επίτροπε δύο λεπτά για να ψηφίσουμε γιατί εγώ δεν έχω ανακοινώσει να σας κάνω. Δεν ξέρω αν έχετε εσεί σχόλια ή προτάσεις για την ημερήσια διάταξη. Όχι. Ωραία. Οπότε πάμε να ψηφίσουμε την θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020. Όπως ξέρετε, στις 29 Νοεμβρίου του 2016 η Ρέτζη υιοθέτησε την γνωμοδότηση με, του κυρίου ε, Φανίστερ Ρόι και τη κυρία Κρέλ για το πρόγραμμα αυτό, στήριξη διευθυντικών μεταρρυθμίσεων, για, με την εντολή ε, έναρξη ε, διαθεσμικών διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν στι στις 11 Ιανουαρίου του 2017. Εγώ σας έκανα μια παρουσίαση των τριμερών διαλόγων στις προηγούμενες συνεδριάσεις μας και μπορώ να σας πω ότι στις 8 Φεβρουαρίου του τρέχοντος υπήρξε μια άτυπη συμφωνία μεταξύ της διαπραγματευτικής ομάδας και του Συμβουλίου. Είναι πολύ καλό το πακέτο. Το Κοινοβούλιο μπόρεσε να εξασφαλίσει τη συμπερίληψη των εταιρικών σχέσεων και της ε, εξέταση από πλευράς Κοινοβουλίου και την συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών εμπλεκόμενων φορέων για την, και τη διαφορά στην διαφάνεια όμως στην εφαρμογή του προγράμματος. Ε, Βεβαίω η οικονομική, η κοινωνική και εδαφική συνοχή επίσης συμπεριλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα και πριν ψηφίσουμε να, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, δεν ξέρω αν οι εισηγητές θέλουν να πούνε κάτι. Α, ο κύριος Βανίστερ, Ένα πολύ σύντομο σχόλιο για αυτή τη συνεργασία που έχουμε και για τη δουλειά που κάνατε εσείς ως πρόεδρος των τριμερών διαλόγων. Αν δείτε την, το πώς ξεκίνησε αυτό το έγγραφο στο Κοινοβούλιο, θα δείτε ότι ήταν πολύ θεωρητική η προσέγγιση που είχαμε, χωρίς να υπάρχει κάποια σύνδεση με την πολιτική συνοχή. Μετά τη δουλειά που κάναμε, και μετά τι διαπραγματεύσει είναι σαφέ ότι οι εταιρικέ σχέσει έχουν ενταχθεί πλέον στο κείμενο, δεν είναι ότι τα κράτη-μέλη που μπορούν να βρουν μόνα του και να υποβάλουν προτάσει από μόνα του για να έχουν στήριξη για τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. αλλά οι εταίροι από τι περιφέρειες και τι πόλει θα πρέπει να, παρέμβουν επίση. Και το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι ότι έχουμε αναγνώριση πλέον του τι κάνει η πολιτική συνοχή ήδη, γιατί γνωρίζουμε ότι τα τρία τέταρτα των ε, συστάσεων αναχώρα ήδη σχετίζονται με τα θέματα που μας απασχολούν, την οικονομική συνοχή, την κοινωνική συνοχή και τα, διάφορα, τα διάφορων ειδών προγράμματα που υπάρχουν. Υπάρχει λοιπόν ένα σαφέ τμήμα που αφιερώνεται σε αυτό στην συμφωνία και ελπίζω ότι θα ψηφίσουμε σήμερα, θα το ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια σύντομα, Ελπίζω να έχουμε ένα λίγο διαφορετικό εργαλείο με μεγαλύτερη, ευρύτερη στήριξη σε σχέση με το τι είχαμε στα χέρια μας όταν ξεκίνησαν αυτές οι συζητήσεις. Η Κωνσταντσα και εγώ δουλέψαμε πολύ πάνω σε αυτό και καταφέραμε να το περάσουμε. Ευχαριστώ και όλους τους σιώδες συγητές για την στήριξή τους. Και ελπίζω βεβαίως ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα και στην ψηφοφορία. Ωραία. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Χρησιμοποιήστε παρακαλώ τις κάρτες σας. Ψηφίζουμε λοιπόν το συμπεφωνημένο κείμενο μετά από τις ε, διαθεσμικές διαπραγματεύσεις ε, στα πλαίσια του κανόνα 69F4 για, την, ε, για τον κανονισμό του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος στήριξης διευθυντικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017-2020. 20. Πολύ μακροσκελής τίτλος. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ναι, να διακόψω προς την ψηφοφορία. Μήπως μπορείτε να ελέγξετε ότι κάθε πολιτική ομάδα έχει τόσο στο αριθμό μελών. Because we have three more votes. Γιατί βλέπω να έχουμε τρεις ψήφους παραπάνω από τον αριθμό των μέλων της Επιτροπής μας. Okay. So we vote again. I'm sorry. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Δεν δουλεύει σωστά το σύστημα ίσως. Για δεύτερη φορά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. το κοινό μας κείμενο. Λοιπόν, το συμπεφωνημένο κείμενο εγκρίνεται. 26 ψήφοι υπέρ και 9 κατά. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές. Περάσαμε λοιπόν το χρόνο ψηφοφοριών, δεν έχουμε άλλες ψηφοφορίες και προχωρούμε στην ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο την κυρία Κρέτσου. Δεν θα εξηγήσω γιατί είσαστε εδώ. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψε και στο παρελθόν και σας δίνω μέσα στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έντιμα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακών Θεμάτων. Καλό απόγευμα. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη εξ αρχής, γιατί δεν μπορώ να μείνω Έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση των, του Σώματος των Επιτρόπων και ελπίζω θα έχετε κατανόηση. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση πάντως να έρθω ενώπιόν σας. Πριν από δύο εβδομάδες, όπως είπε και η Πρόεδρό σας, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την εθνική την ε, πρόταση για τα αντιμετώπιση των καταστροφών και έχουμε το παράδειγμα του σεισμού στην Ιταλία και άλλων φυσικών καταστροφών που έχουν πλήξει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρει και συζητείτε αυτή την πρόταση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι απόλυτα διαθέσιμη για να σας δώσω οποιασδήποτε διευκρινήσεις ώστε να μπορέσει να προχωρήσει ο φάκελος αυτό το ταχύτερο δυνατό. Έτσι με μια ταχεία και αποτελεσματική συνεργασία μπορούμε να επιτύχουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να ευδοκιμήσει αυτή η πρόταση για το, για το Ταμείο για την Αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών και με την πρόταση Omnibus έχουμε και περαιτέρω ευκαιρίες. Εσείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδίω της Επιτροπής Ρέτζι έχετε ήδη από πολύ καιρό ζητήσει να υπάρξει μια απλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομίζω ότι αυτή η πρόταση θα διευκολύνει το έργο όλων μας, παρέχοντας συγχρόνως ένα σταθερό πλαίσιο για αυτούς οι οποίοι λειτουργούν και εφαρμόσουν την πολιτική αυτή επιτοπίως και επίσης θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση θα συνδέσει την περιφερειακή πολιτική με το σχέδιο επενδύσεων ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν περισσότερες περιφέρειες Ευρώπης και να δημιουργηθούν και περισσότερες τοπικές ευκαιρίες επενδύσεων. Βασίζομαι λοιπόν στην εμπειρογνωμοσύνη σας και στην πολιτική σας κρίση, ώστε να διατηρηθεί το πνεύμα της πρότασης και να εξασφαλίσετε ότι οι βελτίωσεις που θέλουν να επιφέρουν να φτάσουν ως τους τελικούς δικαίουχους και είμαι στη διάθεσή σας φυσικά να απαντήσω τα ερωτήματά σας. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, το μέλλον της πολιτικής συνοχής και την επικοινωνία σε σχέση με την πολιτική αυτή. Πρωτού μπούμε στην συζήτηση, θα ήθελα να πω Ό,τι αφορά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την καθυστέρηση της εφαρμογής στην ε, περιφερειακή πολιτική. Καταλαβαίνω τις ανησυχίε σα, Η πολιτική συνοχής είναι ένα από τα βασικά στοιχεία ε, επενδύσεων και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καθυστέρηση σημαίνει καθυστέρηση στην ανάπτυξη, θέσει απασχόληση σε υποδομέ όπω είναι σχολεία και νοσοκομεία. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξουν ταχαίω οι απαραίτητε δράσει, ιδίω στι περιοχέ που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Θέλω να σα διαβεβαιώσω, όπω τόνισε και στην πρόσφατη Ολομέλεια, ότι η πολιτική μα αποδίδει καρπού. <clears throat> Αυτή τη στιγμή 180 δισεκατομμύρια ευρώ, ευρώ έχουν επενδυθεί στην ε, πραγματική οικονομία και έχουμε πάνω από 300 σχέδια που είναι εν εξελίξει στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είμαστε στην ίδια κατάσταση περίπου <clears throat> όπως το χρονικό διάστημα 2007-2013 προχωρούν λοιπόν οι επιλογές των προγραμμάτων και η εφαρμογή των προγραμμάτων. Αυτό είναι που έχει σημασία σε σχέση με την πολιτική αυτή και η ελπίδα μου είναι ότι η επιλογή των προγραμμάτων και η υλοποίησή τους θα αντανακλάται και στην εκταμείευση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύγχρονος φυσικά είναι απαραίτητο να επιταχύνουμε τις διαδικασίες αυτές, όπως είπε και ο κ. Φανίς Φλερόι στην συζήτηση της Ολομέλειας και όπως είπατε πολλοί από εσά, εμείς συνεργαζόμαστε με όλα τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες ιδίως εκεί που έχουμε εντοπίσει ιδιαίτερα σημεία συμφόρησης. Κοιτάζουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα στο επόμενο πλαίσιο χρηματοδότησης. Υπάρχουν οι προσπάθειες μας για την απλοποίηση και πιστεύω ότι θα αποφέρουν καρπούς και έρχομαι και στο δεύτερο σημείο που θέλω να δείξω σήμερα το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής Η Κέρστιν Βάστφαλ εργάζεται, πρώην συνάδελφός μου, εργάζεται στο θέμα αυτό και πιστεύω ότι το συμπέρασμα από αυτή την εργασία είναι ότι χρειαζόμαστε για το μέλλον μια στεναρή πολιτική συνοχή και επίση να δώσουμε ένα σαφέ πολιτικό μήνυμα από τώρα ότι μετά από το δημοπίσμα του Brexit και την εκλογή του Donald Trump έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικές εκλογές στις κάτω χώρες, στην Γαλλία και την Γερμανία και επομένως πρέπει να δώσουμε μια πιο πολιτική χρειά σε όλα αυτά. Πρέπει να δώσουμε ένα πολιτικό σαφές μήνυμα στους 20 τα 20 εκατομμύρια Ευρωπαίων που είναι άνεργοι, στα 100 εκατομμύρια Ευρωπαίων που είναι κάτω από το κατόφλι της ένδυας, ότι το μέλλον τους δεν βρίσκεται στο λαϊκισμό, δεν βρίσκεται στην επιστροφή στο παρελθόν. Εγώ προσπαθώ να τονίζω όπου πηγαίνω ότι νοιάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η πολιτική συνοχή βελτιώνει την καθημερινή ζωή των πολιτών και δίνει ευκαιρίε σε όλου. Πράγματι, αυτό είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα για την πολιτική συνοχή. Είμαι πεπισμένη ότι αυτή είναι ακριβώς η πολιτική συνοχή που περιμένουν από εμά οι πολίτες μας και η πολιτική η οποία αντιμετωπίζει πραγματικές προκλήσεις, τη δημιουργία καινοτομίας και νέων δεξιοτήτων, αντιμετώπιση της ένδυας, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές της Ευρώπης, όσο ανεπτυγμένες και να είναι. Είναι απαραίτητη λοιπόν η πολιτική συνοχή για όλε τι περιοχέ τη Ευρώπη, γιατί με τον τρόπο αυτό δίνει σε όλε τι περιοχέ τη Ευρώπη τη δυνατότητα να παίξουν το ρόλο του σε ό,τι αφορά την επίτευξη των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιε περιοχέ απ' έξω. Για όλου αυτού του λόγου όμω είμαι πεπισμένη και για δύο ακόμα στοιχεία τη πολιτική συνοχή, ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι επενδύσει μα βρίσκονται στην ε, καρδιά της του Ευρωπαϊκού Θεματολόγιου Μεταρρύθμισης και ότι θα μπορέσουμε να έχουμε εξοικονομήσεις και αποτελεσματική διαχείριση και αλλαγέ όπου αυτό είναι απαραίτητο. Και επιπλέον θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πολιτικές μας και είμαι σίγουρη μπορούμε να βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ του να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και συγχρόνως να έχουμε αποτελέσματα για τη συνοχή, για την απασχόληση και την οικονομική μεγέθυνση. Δεν θα επεκταθώ τώρα περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και κάποιες περαιτέρω συναντήσεις για τα θέματα του τι θα γίνει πέραν του 2020. Αύριο θα είμαι στην Βασοβία για στη συνδιάσκεψη θα εξετάσει το τι θα γίνει μετά το 2020. Τον Ιούνιο θα έχουμε και ένα φόρμα για τα θέματα αυτά και έτσι θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες πολιτικές. Ξέρετε όπως και εγώ ότι οι συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων είναι απαράγραπτες, αλλά δεν είναι ικανές για να αλλάξουν από μόνες τους την ροή της ιστορίας. Θα πρέπει οι πολίτες να μας υποστηρίξουν. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι πολλοί από τους πολίτες μας δεν έχουν ακούσει ποτέ ότι υπάρχει πολιτική συνοχή. Είναι κοινό μας καθήκον να το τροποποιήσουμε αυτό. Προσπαθούμε με φορεί επικοινωνία στα κράτη-μέλη και τι περιφέρειε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε ξεκινήσει μια εκστατεία που έχει τίτλο Η Ευρώπη, η περιφέρειά μου, ώστε να δείξει στους πολίτες τι γίνεται και να αναζητήσει εταίρους επιτοπίως και προφανώς μπορείτε και εσείς να συνεισφέρετε ιδέες. Εγώ που πηγαίνω προσπαθώ να επισκεφθώ τα διάφορα σχέδια και προγράμματα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών εκεί και θα παρουσιάσουμε την άνοιξη αργότερα ένα σχέδιο δράσης Ξέρετε ότι η επικοινωνία είναι από τα κύρια μελήματά μου αυτή τη χρονιά, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την πολιτική μας και να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Είμαι σίγουρη ότι μπορώ να βασιστώ και στη δική σας υποστήριξη για όλα αυτά τα εγχειρήματα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, ευχαριστώ. Ως ήθιστε θα ξεκινήσει ο πρώτος γύρος ε, ερωτήσεων. Θα ακούσουμε ερωτήσεις και σχόλια των συντονιστών. Ο κύριος Βανίστελ Ροϊ Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο που παρίσταται και μας δίνει τη δυνατότητα να θέσουμε κάποια σημαντικά σημεία. Ευχαριστώ που ήσασταν τόσο συγκεκριμένοι σήμερα, διότι επαναλάβατε την πρότασή σας να υποβάλλετε ένα σχέδιο δράσης για την επικοινωνία. Είναι σημαντικότατο αυτές τις ημέρες. Να δείξουμε τι κάνουμε δεν είναι μόνο θέμα γενικό, αλλά αφορά τις πόλεις και τις περιφερειές μας. Και νομίζω ότι πολλοί πολίτες στην Ευρώπη είναι πρόθυμοι να μιλήσουν γι' αυτό. Θέλουν να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις και ιστορίες. Και μια περίοδο λαϊκισμού πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δεύτερον, χαίρομαι που αναφερθήκατε στο μέλλον. Εν τη αυτή περίπτωση, με την επικείμενη λευκή βίβλο, που θα ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα το μέλλον της Ευρώπης. Ότι χρειάζεται τώρα συνοχή παραπάνω από ποτέ. Χρειάζονται διαθετικές πολιτικές, περισσότερο από, πολλές. από ποτέ. Συγγνώμη. Και θα πρέπει να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας. Είναι σαν να ομφαλοσκοπούμε τώρα. Βασικά είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για να κρατήσουμε ενωμένη την Ευρώπη. Διότι υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες στην Ευρώπη ήδη σήμερα. Κάποιοι κινούνται ταχύτερα από άλλου. Αλλά αν συμφωνήσουμε επί κοινού θεματολογίου, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλουμε να συμφωνήσουμε, χρειάζεται να έχουμε μια βάση. Και αυτή είναι η πολιτική συνοχής. Και σε συνδυασμό με τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που έχουμε στη διάθεσή μας, όχι μόνο με τα ρυθμιστικά προγράμματα και το πρόγραμμα για την υποστήριξη των διαφόρων διαθωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και η πολιτική συνοχή, όπω η ρεσιμότητα εκ των υστέρων, προπολογισμό βάσει επιδόσεων, ο τρόπο προετοιμασία και συνέχεια που θα δοθεί. Όλα αυτά είναι σημαντικά για όλη την Ευρώπη. Και πιθανότατα σε συνδυασμό με αυτά που πετύχαμε με τις προσεγγίσεις ευφυής, ευφυούς εξειδικεύσεως, όχι απλώς να κατασκευάζουμε σχολεία και να κατασκευάσουμε δρόμους και κοινωνικά προγράμματα, αλλά να διασυνδέουμε εκείνους που είναι στην πρώτη γραμμή ε, και μπορούν να ακολουθήσουν έτσι οι άλλοι. Δεν μπορούν όλοι να παράγουν τα ίδια προϊόντα στην οικονομία τους. Έτσι δημιουργείται κάτωθεν προσέγγιση που πλησιάζει και το θεματολόγιο με βάση τη γνώση. Θεματολόγιο στο οποίο βασιζόμαστε για την επόμενη 20 ετία στην Ευρώπη. Αφορά τους πόρους μας, τους λαούς μας. Η σημερινή ομιλία της Επιτρόπου με βοήθησε να πω ότι ναι, πράγματι πρέπει να βελτίσουμε την ορατότητά μας. Όλοι μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του συναδέλφους να δείξουμε ότι η συνοχή είναι από τους βασικούς στόχους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020 με 27 χώρες. Εντάξει, μου δημιουργήσατε την κατάλληλη ατμόσφαιρα για τη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Κρέολ. Κύριε Κοτσολίν. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Καθορίσατε λοιπόν ότι χρειάζεται ενισχυμένη επικοδομητική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πάνω απ' όλο πιστεύω ότι έχουμε χρόνο για να εμπλεχθούν και οι πρωταγωνιστές της πολιτικής συνοχής. Πιστεύω ότι μια από τις επιλογές που θα πρέπει να κάνουμε και σαν Κοινοβούλιο και σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χάρη στη δημιουργία ενός φόρουμ τον Ιούνιο ε, στόχος μας είναι να συμμετάσχουν οι περισσότεροι φορεί τη πολιτική συνοχή. Δεν πρέπει να κλειστούμε εμεί στι Βρυξέλλε και να συζητούμε μεταξύ μα. Χρειαζόμαστε θετικέ επαφέ και σχέσει με τι περιφέρειες, τις κοινότητες, τις πόλεις, τις οργανώσεις του κόσμου τη εργασία, του εθελοντέ. Θέλουμε να έχουμε δυνατότητα να ακούμε και να πρωταγωνιστήσει η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών. Η πολιτική συνοχή πραγματικά από τι πρώτε κινήσει τη μεταρρύθμισης να γίνει ένα μεγάλο εργαλείο επικοινωνία, κοινωνικής επικοινωνίας. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πρώτο σημείο. Πάνω σε αυτό θα πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία όλοι μαζί. Ότως ώστε να έχουμε μέγιστη συμμετοχή όλων των αρχών, όλων των δυνάμεων και μετά συγκεκριμένα αυτοί θα ασκούν την πολιτική συνοχή. Δεύτερο θέμα. Αν επιλέξουμε το δρόμο της ενισχύσεως μέσω καινοτομίας αλλά να ενισχύσουμε και να παγιώσουμε την πολιτική συνοχή σαν κάτι στατηγικό τα επόμενα χρόνια. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Από εκεί απορρέουν διάφορε επιλογέ, ξεκινώντα τον προπολογισμό, του πόρου που θα δεσμεύσουμε και θα διθέσουμε. Πρέπει πάνω απ' όλα να επιλέξουμε αυτή τη γραμμή, τη βασική γραμμή που θα ακολουθήσουμε. Αν η πολιτική συνοχή πρέπει να είναι η πολιτική των επόμενων ετών τη Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ναι. Πρέπει να δώσουμε θετική απάντηση σε αυτό το ερωτηματικό, να προσπαθήσουμε παρόλες τις διαφορές και αποκλήσεις απόψεων που υπάρχουν μεταξύ μας και μεταξύ χωρών και μεταξύ τοπικών κοινοτήτων, παρόλα αυτά να δώσουμε ένα μήνυμα προς την Ευρώπη ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε τη δικασία τη μεταρρύθμιση τη πολιτική συνοχή και θέλουμε να ενισχύσουμε την πολιτική συνοχή του τρόπο, να την παρασπιστούμε, διότι γνωρίζουμε ότι αυτά είναι από τα ελάχιστα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα ούτω ώστε να εφαρμόσουμε επενδυτικέ πολιτικέ, αναπτυξιακέ πολιτικέ στην Ευρώπη. Και μετά θέλουμε να λύσουμε και κάποιου, κάποια προβλήματα. Εντάχει θα αναφέρω κάποιου από τους, τους κόμπους που έχουμε να διαλύσουμε και να λύσουμε. Ε, μετά λοιπόν από τα σχεδόν 8-9 χρόνια της κρίσης που έχουμε στην πλάτη μας, κάποια σημεία θα πρέπει να επιληθούν οριστικά και η σχέση μεταξύ πολιτικής συνοχής, δηλαδή της ανάκαμψης των δημοσίων επενδύσεων και της οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να εξεταστεί. Τα προγράμματα εξυγίανσης που εφαρμόζουν τα διάφορα Τι είδους σχέσεις πρέπει να έχουν όλα αυτά μεταξύ τους. Καμιά φορά, χωρίς να λαμβάνουμε πλήρως υπόψη, παρά τη μεγάλη τεκμηρίωση, όταν εφαρμόζουμε λιτότητα, εξυγίανση και συστολικές αυτές ε, πολιτικές ε, δεν πετυχαίνουμε την σωστή εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, να μειωθούν οι αποστάσεις οι κοινωνικές, οι εδαφικές και οι περιφερειακές. Ε, πολύ συχνά ήταν το μόνο εργαλείο που έχουμε στη θέση μα η πολιτική συνοχή. Και τώρα ήρθε η στιγμή πάνω σε αυτό να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Να δούμε πώ μπορούμε να προωθήσουμε την πολιτική συνοχή, να περάσει τη νέα φάση η πολιτική συνοχή και πώ σχετίζεται με την οικονομική διακυβέρνηση. Δεύτερο μεγάλο ζήτημα λοιπόν που γεννάται από το νέο κοινοβούλιο με αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το θέμα αυτό. Σχέσεις μεταξύ επενδυτικών σχεδίων του, του σχεδίου Juncker και της πολιτικής συνοχής. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε και να εκφραστούμε σαφώς στη συζήτηση. Να, αν είναι αυτή η επιλογή, τι σημαίνει, τι συνεπάγεται αυτή η επιλογή όσον αφορά την πολιτική συνοχή, τι συνεπάγεται αυτή η επιλογή όσον αφορά το σχέδιο το Juncker. Συγκεκριμένα, τι συνεπάγεται όσον αφορά την εργοποίηση των διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων. Τέλος, το μεγάλο ζήτημα, πάνω στο οποίο συχνά στρέφουμε την προσοχή μας. Ανεφερόμαστε στα 20 εκατομμύρια στους νέους, τους ανέργους. Πώς τους μιλάμε. Πώς η πολιτική συνοχή μπορεί να μιλήσει σε αυτούς τους ανέργους νέους. Στην προηγούμενη θητεία μαζί με τις περιφέρειες κάναμε επιχείρηση διεύρυνσης του φάσματος των ε, περιοχών που συμμετέχουν στην πολιτική συνοχή. Ενεπλέκονται περισσότερε περιφέρειες στην πολιτική συνοχή. Το συζητήσαμε εκτενώ. Ήταν με επιλογή αποφασιστική αυτή που έγινε. Διότι δημιουργήσαμε ευρύτερη συμμαχία όσον αφορά την πολιτική συνοχή. Αυτό πράγματι ήταν κάτι θετικό σαν αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι παρόμοιο όσον αφορά τις νέες γενιές των Ευρωπαίων. Δηλαδή αυτή τη φορά το θέμα είναι πώς η πολιτική της συνοχής γίνεται ένας ενδεχόμενος σύνοχο, ε, σύμμαχος των νέων ανθρώπων. Να εξυπηρετήσουμε αυτές τις νέες γενιές, να τις βοηθήσουμε ώστε να διαθέσουν το ταλέντο τους ε, για την Ευρώπη του μέλλοντος. Ε, ε, είναι μια μεγάλος, ένας μεγάλος παράγον κοινωνικός στην πολιτική συνοχή. Και αυτό αφορά το ζήτημα που συζητούμε εκτενώς. Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να παρουσιάσουμε την πολιτική συνοχή. Είναι παράδοξο. Καμιά φορά κάνουμε πολύ σημαντικά, σημαντικότατα πράγματα και δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό Πώς αλλάζει μια πολιτική ή μια τοπική κοινότητα, μια πόλη από τη χρήση κοινοτικών πόρων. Ήρθε η στιγμή ίσως να το τονίσουμε αυτό. Να μην το θέσουμε σε θέμα προπαγάνδας ή επικοινωνίας. Αλλά πώς δημιουργούμε πολιτικές που δημιουργούν κάνουν τους κοινωνικούς φορείς να αισθάνονται ότι ωφελούνται από την πολιτική συνοχή. Ίσως κάποιες πτυχές είναι αυτές ε, τη συζήτηση που ξεκινήσει για την αναθεώρηση της πολιτικής συνοχής τους επόμενους μήνες αυτό το χρόνο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Τόμασιτς. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Δεν είναι αρκετό να λέμε στους ανθρώπους στα κράτη-μέλη ότι έχετε διάφορα κονδύλια στα διάφορα ταμεία και από εσά εξαρτάται να υπάρχουν μάλλον κάποια κονδύλια σε διάφορα ταμεία και πώς σας κρατάτε να μάθετε πώς θα τα πάρετε. Νομίζω ότι κάποιοι που μπορούσαν να ε, απασχολήσουν 200 ανθρώπους ή παραπάνω, γιατί ε, ε, πολλές φορές τα παράτησαν γιατί δεν υπήρχε διαφάνεια. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια από τα ταμεία αυτά με έναν απλό τρόπο. Το θέμα δεν είναι να τους πούμε «Να, εδώ είναι τα κονδύλια», βρείτε τώρα εσείς τον τρόπο να, να τα πάρετε. Γιατί κάποιοι μπορούν να το κάνουν αυτό εύκολα και εκμεταλλεύονται το σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη σίγουρα θα μπορέσουν να συνεργαστούν με διαφανή τρόπο από την αρχή ως το τέλος, γιατί είναι και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιες περιπτώσεις απατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω την κυρία Επίτροπο και θα ξεκινήσω με κάποια σχόλια και κάποια ερωτήματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι μας θέλουμε να συνεχιστεί ε, να συνεχίσει την επιτυχία της η πολιτική συνοχής και στην ε, πρωτολογία σας ε, κύριε Επίτροπε είπατε ότι θέλετε να το υποστηρίξετε αυτό, να το προωθήσετε και θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν ώστε η πολιτική συνοχής να συνεχιστεί και να δείξει τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της αλληλεγγύης. Σίγουρα τους επόμενους μήνες, τα επόμενα ένα-δύο χρόνια θα υπάρξουν πολλές προσπάθειες να υπάρξει μείωση των, της για την πολιτική συνοχή. Και αυτό μπορεί να έχει σχέση και με, την, με το νέο σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση δηλαδή του ρόλου των περιφερειών και των πόλεων. Ξέρω ότι στις 5 έχετε την έκτακτη αυτή συνεδρίαση του Κολεγίου των Επιτρόπων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε ίσως να έχετε πιο συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις για μένα μετά από αυτή τη συνεδρίαση. Αλλά θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο ρόλος που θεωρεί η Κομισιόν ότι έχουν να παίξουν οι πόλεις, οι περιφέρειες και όλες οι διάφορες δομές που είναι όμως απαραίτητες για να υπάρχει μια σωστή και ποιοτική πολιτική συνοχή έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα κονδύλια δαπανώνται με το σωστό τρόπο. Γιατί ε, το μεγάλο κομμάτι των κονδυλίων περνάει από τις περιφέρειες και τις πόλεις. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε εσείς πώς βλέπετε, ποιος, είναι, ποιος βλέπετε να είναι ο ρόλος των πόλεων και των περιφερειών στο μέλλον και τι πιστεύει η Κομισιόν του κυρίου Γιούνκερ από αυτού, ο κύριος Παπαδημούλης. Ε, κυρία Επίτροπε, η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής του Ευρωκοινοβουλίου θέλει οπωσδήποτε στην πολύ μεγάλη της πλειοψηφία οι πολιτικές συνοχής να ενισχυθούν και να γίνουν πιο αποτελεσματικές για τη μείωση των ανισοτήτων και των περιφερειακών και των κοινωνικών που οι ίδιες οι στατιστικές της Eurostat και της Κομισιόν δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μεγαλώσει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και μέσα στην Κομισιόν η δική σας βούληση για να έχουμε ισχυρές πολιτικές συνοχής βρίσκει καμιά φορά εμπόδια. Και κονδύλια υπέρ των πολιτικών συνοχής αντί να ενισχυθούν, μειώνονται προκειμένου να καλυφθούν άλλες ανάγκες. Επομένως, η ερώτησή μου είναι γιατί πρέπει τα έκτακα κονδύλια για την αντιμετώπιση των αναγκών που απορρέουν από την προσφυγική κρίση να αφαιρούνται από τα κονδύλια των πολιτικών συνοχής και όχι από κάπου αλλού. Και η δεύτερη ερώτηση που αφορά ειδικότερα στη χώρα μου την Ελλάδα. Και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν συμφωνήσει σε κάποιους στόχους σε ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης με ευθύνη όχι τόσο τη Κομισιόν όσο συγκεκριμένων κρατών μελών η υλοποίηση αυτού του προγράμματο του συμφωνημένου βρίσκεται σε ποσοστό 5% και κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία σηκώνουν με ελλειπή αλληλεγγύη το βάρος αυτής της προσφυγικής κρίσης. Τι μπορεί παραπάνω να κάνει η Κομισιόν και πώς μπορεί παραπάνω να πιέσει διάφορα κράτη-μέλη έτσι ώστε η αλληλεγγύη ω λέξη στο θέμα αυτό να μην είναι ένα γράμμα κενό. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, που είσαστε στη διάθεσή μας σήμερα. Ευχαριστώ και για την πρωτολογία σας. Συμμερίζομαι όλα όσα είπατε για την ε, σημασία της πολιτικής συνοχής. Είναι όντως ένα σύμβολο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά ε, και η ε, αλληλεγγύη είναι ένα καλό εργαλείο για τους ε, πολίτες της ε, Ένωσης ε, έτσι ώστε να υπάρχουν κοινέ αρχές για όλους τους πολίτες τις οποίες θα πρέπει να τηρούν. Το ερώτημά μου είναι σαφές γιατί μιλήσατε και για το Omnibus. Πώς θέλετε να εξασφαλίσετε ότι θα προχωρήσει με επαρκώς επικοδομητικό τρόπο η πολιτική συνοχής ε, και τι θα γίνει με, την, ε, ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή από τα άλλα ταμεία, η μεταφορά των κονδυλίων, πώς θα γίνει σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες όμως έχουν άλλο τελείως στόχο και άλλες κατευθυντήρες γραμμές και άλλες αρχές. Πώς θέλετε να εξασφαλίσετε την συνέχεια της ε, πολιτικής συνοχής ε, ας πούμε για διάφορους τομείς από καθημερινά πράγματα μέχρι μεγάλους στόχους όπως την ε, κλιματική αλλαγή. Ξέρω ότι σε αυτό σας απασχολεί ιδιαίτερα και ακριβώς λόγω αυτού του υποβάθρου έχουμε και εμείς κάποιες ανησυχίες ότι αν, έχουμε αυτό το, αν δούμε το Ταμείο για τις ε, Σταδικές Επενδύσεις εκεί υπάρχει πολύ μικρή ε, κοινωνική διάσταση και το 4% μόνο των κονδυλίων πηγαίνουν εκεί που πρέπει, στην πολιτική συνοχή δηλαδή. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε συζητήσουμε ε, πώς θα προχωρήσει η πολιτική συνοχή, πώ θα χρηματοδοτείτε και στο μέλλον πώ θέλετε εσεί να το ε, πραγματοποιήσετε αυτό. Γιατί μιλούμε για ε, δυνατότητες μεταφοράς κονδυλίων προς, την, προς τα διάφορα, από τα διάφορα ταμεία για την πολιτική συνοχή. Ένα δεύτερο ερώτημα που έχω να κάνω είναι για το μετά το 2020. Μήπως μπορείτε να μας πείτε λεπτομερέστερα τι γίνεται σε ό,τι αφορά τις ε, για, τις εκ ε, για την εκτονιστέρων των υστέρων αιρεσιμότητα. Και το τελευταίο ερώτημα που πάντα θέτω, γιατί είναι σημαντικό για μας, τι γίνεται με τις εργασίες στην Κομισιόν σε ό,τι αφορά <coughs> το GDP and beyond, την ε, περαιτέρω δηλαδή εξέλιξη του ΑΕΠ, μια που τώρα έχουμε πολλές ε, εξελίξεις με, τις, ε, με την ε, ισοτιμία σε ό,τι αφορά την κατανομή των ε, κονδυλίων, με τους προϋπολογισμούς. Εσείς πώς, πώς βλέπετε να προχωρά αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που γίνονται και από άλλους επιτρόπους. Πείτε μας και εσείς τη δική σας άποψη. Κυρία Ντεμάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, στις 30 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο όπου περιέγραφε λεπτομερώς τις προσαρμογές τεχνικής φύση, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάποια κράτη-μέλη. Βάσει των υπολογισμών, η Ιταλία θα είχε δικαίωμα σε 1,6 δις. Αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να πάνε ε, για την καταπολέμηση ενεργεία των νέων, για την κρίση μεταναστευτικό και για επενδύσει μέσω χρηματοστικών ε, μέσων, δηλαδή συνέργεια μεταξύ των Διευθυντικών Ταμείων και του σχεδίου Juncker. Εσεί ανακοινώσατε κατά τη διάρκεια τη επίσκεψη στην Ιταλία ότι περίπου 200 εκατομμύρια από αυτό το 1,6 δι προοριζόταν από την Ιταλική κυβέρνηση για την ανοικοδόμηση μετά του ε, σεισμού. Γνωρίζουμε όμω, όπω είπατε κι εσεί, ότι οι διαπραγματεύσει με τι κυβερνήσει, άρα και με την Ιταλική κυβέρνηση, ακόμα συνεχίζονται με τις κυβερνήσεις που δέχονται συμπληρωματικούς πόρους ε, στα πλαίσια της τεχνικής προσαρμογής. Λοιπόν, θα ήθελα να γνωρίζω, αν μπορείτε να μας πείτε, αν αυτό είναι ορθό. Θα ήθελα να ξέρω ποια ήταν τα περιθώρια λιγμών από το 1,6 δις. Υπάρχει δυνατότητα από πλευρά κρατών μελών ε, να διαθέσουν με διαφορετικό τρόπο τα χρήματα και στη συγκεκριμένη περίπτωση Ιταλίας θα έχει τη δυνατότητα η χώρα να δώσει περισσότερα χρήματα από τα 200 εκατομμύρια για την ανοικοδόμηση μετά τους σεισμούς. Πάντα αν η χώρα ζητήσει κάτι τέτοιο. Τελευταία ερώτηση, διότι δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν αυτές οι προσαρμογές είναι πάντα, οι, αν υπόκειται στη χρηματοδότηση. Και αν ναι, επαναλαμβάνω ότι εν τη αυτή περιπτώση δεν κατανοήσαμε πόσο σημαντικές είναι οι δημόσιες επενδύσεις σε μια περίοδο κρίσης και συνεπώς αυτές οι επενδύσεις όπως αποφασίστηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο στο ψήφισμα που ενεκρίθη με πλειοψηφία, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον υπολογισμό του ελλείμματος. Ευχαριστώ. Ο κ. Μπλουά είναι ο τελευταίος που λαμβάνει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, άκουσα με μεγάλη προσοχή τα λεγόμενά σας, τη δήλωσή σας και πιστεύω ότι δυστυχώς παραμένετε πάντα ίδια δυστυχώς. Εγώ σημείωσα ότι σε κανένα <clears throat> σημείο της ε, δήλωσής σας δεν θέλετε να διαμφισβητήσετε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πηγαίνετε προς τον τοίχο κατευθείαν επιταχύνοντας και χτυπάτε και την κόρνα. Νομίζω ότι δεν ακούτε την άποψη των πολιτών, των λαών. Δεν βλέπετε αυτά τα 20 εκατομμύρια που είναι άνεργοι, τα 9 εκατομμύρια των Γάλλων που είναι τα θύματα της πολιτικής που ακολουθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, οδηγία των ε, αποσπασμένων εργαζομένων με τις μαζικές μετακινήσεις επιχειρήσεων στη δική μου ε, περιοχή υπάρχει μια επιχείρηση πολύ γνωστή, η Whirlpool, η οποία θα μετακινηθεί στην Πολωνία όπου μπορεί να εκμεταλλευτεί εργαζόμενους με μικρότερο κόστος. Και αυτό γίνεται δυνατό λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εσείς, κυρία Επίτροπε, δεν θέλετε να αμφισβητήσετε τίποτα. Λέτε όλα δεν είναι καλώς. Όλα πάνε πολύ καλά. Τι έχετε λοιπόν να πείτε, μονάχα να επικρίνετε την ψήφο των Βρετανών για τον Brexit. Μα είναι δική του επιλογή. Την εκλογή του Τραμπ, μα είναι υπόθεση των Αμερικανών. Έχετε στραφεί εναντίον αυτού που ονομάζεται λαϊκισμό. Εγώ όμως είμαι υπερήφανος που είμαι λαϊκιστής γιατί ο λαϊκιστής είναι αυτός ο οποίος ακούει τη φωνή των λαών. Και δεν μιλήσατε καθόλου και για την Αυστρία, όπου οι λεγόμενες λαϊκιστικές δυνάμεις φτάσανε το 47% στις προεδρικές εκλογές. Δεν μιλήσατε και για το λαϊκισμό στην Ιταλία, γιατί το δημοψήφισμα που υποστήριξε η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκόμισε ένα μεγάλο ράπισμα ή για την Ουγγαρία, όπου 96% του ουγγρικού λαού ψήφισε υπέρ της υποδοχής των μεταναστών. Και φυσικά δεν είπατε τίποτα για τις ε, μελλοντικέ εκλογές στις κατοχώρες, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Μα κυρία Επίτροπε, περιμένετε και πάλι να έχετε σημαντικούς κλειδονισμούς. Θα πρέπει να τους περιμένετε. Ξέρω δεν σας αρέσει λέτε ότι θέλετε να επικοινωνήσετε περισσότερα, αλλά αν η ανακοίνωσή σας είναι το να κρίνετε φυλάδια όπως αυτό εδώ για να προωθείτε την υποδοχή των μεταναστών σε όλες τις ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως σε τομείς που υποτίθεται ότι είναι η αγροτική ανάπτυξη, να ξέρετε ότι την επόμενη φορά θα σας αρρώσει η λαϊκή ψήφος. Και εάν πάλι θέλετε να τονίζετε την ε, ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πάτε στράφη. Αυτό ήταν δήλωση, δεν ήταν ακριβώς ερώτηση. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση που θέλουμε να, διαμυ... να διαμυφθεί τώρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλα τα ερωτήματά σας και τη δήλωση που ακούστηκε τώρα και η κυρία Επίτροπος έχει τώρα το λόγο για να δώσει κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις συνεισφορές σας. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα που άκουσα όλες αυτές τις απόψεις που διατυπώσατε. Μου λείπουν οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Βανίστλεροι έθεσε ένα ερώτημα σε σχέση με το οποίο νομίζω ότι πράγματι μπορεί να διαιωνίσουμε τα ίδια σφάλματα. Όταν εγώ ήμουνα εδώ παρατηρήτρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση για τον λαϊκισμό. Αλλά τώρα δεν λέγαμε τότε τι είχε επιτύχει η ευρωπαϊκή πολιτική με τα χρόνια. Αφήναμε να προχωρεί το έργο μας και με τον τρόπο αυτό γινόταν αξιόπιστο, αλλά δεν είχαμε αρκετή επικοινωνία σε σχέση με τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής. Γι' αυτό βλέπω ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο του ρόλου μου και μια προτεραιότητά μου για φέτος είναι η επικοινωνία. Ο Κάλλος Μουέντας που ήταν ο αρμόδιος για τα θέματα έρευνας και ε, που είναι αρμόδιος για τα θέματα έρευνας και ανάπτυξης και ήταν στο Μάντσεστερ το καλοκαίρι, μου είπε ότι θα πάει στο Πανεπιστήμιο της Μαχαιστρίας για να παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα και εμείς γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο αυτό έχει επιδοτηθεί με 250 εκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και λέμε επομένως σαφώς ότι εμείς συνεισφέρουμε. Από την άλλη μεριά ο Κάρλος δεν είδε κανένα ίχνος της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρώτησε τον ε, τώρα του Πανεπιστημίου, αν, γιατί δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ίχνος της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου του, του είπαν ότι απαγορεύεται να θέτουν την Ευρωπαϊκή Σημαία σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Δεν είναι λοιπόν η μόνη τέτοια περίπτωση που ο τοπικός δήμαρχος παίρνει όλα τα θετικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν δείχνει ότι προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό έχουμε ένα σχέδιο την επικοινωνία. Ξέρετε ότι τα κρατημέλη ήδη μπορούν να βασιστούν στην τεχνική αρρωγή και να πάρουν τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να χρηματοδοτήσουν δράσεις επικοινωνίας. Αλλά εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα πεπισμένη ότι τέτοιου είδους δραστηριότητε έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να διαφωτίσουμε τους πολίτες για την πολιτική συνοχή. Και να τονίσουμε ότι είναι κοινό μας μέλημα να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ευρύτερη γνώση και ότι οι πολιτικοί όλων των κομμάτων να μπορούν να τονίσουν τον θετικό αντίκτυπο αυτής της πολιτικής στη ζωή των πολιτών. Εδώ η, η περιφέρεια έχει ένα ευρύ τομέα αρμοδιοτήτων. Εγώ ήμουν προηγουμένω στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, όπου συζητήσαμε το ποσοστό σφαλμάτων στην περιφερειακή πολιτική. Αν όμως μια χώρα έχει μόνο 5% ποσοστό μη απορρόφηση, τα άλλα 95% είναι απορρόφηση. Και αυτό είναι επιτυχία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ακούσουμε αυτά που λέει και το ελεκτικό συνέδριο Ξέρουμε όλοι πόσο πολύπλοκη είναι η πολιτική περιφερειακών θεμάτων. Ακούμε συνέχεια αυτή τη ρεδοδοτική που στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η πολιτική συνοχής. Μετά από το 2020 σας τόνισα ποιοι είναι οι στόχοι μου. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τη συζήτηση και απαντώντας τον κύριο Βανίστρερο και στον κύριο Γιάκοβιτς για τη συζήτηση που διαλαμβάνεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση και για μένα είναι σαφές ότι πρέπει να κρατήσουμε ενωμένη την Ευρώπη. Η πολιτική συνοχή πρέπει να καλύψει όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Με ρώτησε ένας Γερμανός δημοσιογράφος γιατί ο προϋπολογισμός δεν περιορίζεται μονάχα στις πιο φτωχές χώρες αφού μειώνεται ο προϋπολογισμός της συνοχής. Για μένα αυτό είναι λάθος γιατί η πολιτική συνοχή αφορούσε από την αρχή όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να καλύψει το χάσμα μεταξύ των φτωχότερων και των πλουσιότερων περιοχών, αλλά επίσης να βοηθήσει τις πλούσιες περιοχές να διατηρήσουν το επίπεδό τους. Όλα αυτά που είπατε λοιπόν κύριε Φανιστερόι για την πολιτική συνοχής που έχετε υποστηρίξει και εσείς ως συνομοθέτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η εκ των προτέρων ερεσιμότητα, η εξειδίκευση, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να βασιστούμε στα ισχυρά σημεία κάθε περιφέρειας και η συνδιάσκεψη που θα γίνει στο Ελσίνκι θα τονίσει αυτά τα σημεία. Η πολιτική συνοχή λοιπόν είναι απαραίτητη για να δώσει σε όλε τι περιφέρειες τη Ευρωπαϊκής Ένωση να προχωρήσουν στη βιομηχανική, ενεργειακή και τεχνολογική μεταλλαγή που διερχόμαστε και είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε και τι ευκαιρίε για όλου του πολίτε παντού να προχωρήσουν προ την κατεύθυνση αυτή. Λυπάμαι που οι περισσότεροι από εμά δεν βλέπουμε αυτά που έχουν γίνει σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Τι δείχνουν τα αριθμητικά στοιχεία, πόσες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί, πόσοι οφείλουν τη θέση απασχόλησής τους στο, στα ευρωπαϊκά σχέδια και τα ευρωπαϊκά ταμεία. Είναι πολύ σημαντικό να μην υπολείπονται κάποιοι από τους πολίτες μας επειδή κάποιος ζήτησε να υπάρχει περισσότερη υποστήριξη των κοινωνικών αλλαγών, της κοινωνικής διάστασης. Πρέπει πράγματι να βελτιώσουμε τον κοινωνικό πυλώνα. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε και τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης, γιατί είναι γεγονός ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο όλες οι περιφέρειες. Είναι διαφορετικό να χρησιμοποιεί κανείς τα περιφερειακά ταμεία για πλούσιες περιοχές των κάτω χωρών και σε φτωχές περιοχές που έχουμε στη Λιθουανία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα με ανοιχτό πνεύμα και να βρούμε τη σωστή διαφοροποίηση ώστε κανείς να μην ενοχλείται, αλλά φυσικά να αποδεχθούμε το ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης και υπάρχουν ιστορικοί λόγοι για αυτές τις αποκλήσεις. Και φυσικά οι ιστορικοί θα μπορούσαν και μόνο να αποφασίσουν τι θα είχε γίνει αν είχαν χρησιμοποιήσει όλες οι χώρες μας τα κονδύλια αυτά από την αρχή. Νομίζω κύριε Κοτσολίνο ότι η συζήτηση που έγινε με τις περιφέρειες της Νότιας Ιταλίας ήταν πολύ επωφελής. Η Ιταλία δεν είναι καινούριο κράτος μέλος αλλά και άλλες χώρες όπως είναι ε, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία που έχουν θυγεί από την κρίση και αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν πρέπει να περιοριστεί η βοήθεια μονάχα στις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι έδωσε ένα σαφές μήνυμα και σας το ξαναλέω ότι χρειαζόμαστε την πολιτική συνοχή περισσότερο από ό,τι ποτέ. Ε, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να περιοριστούμε μονάχα στο status quo. Θα πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής είναι μια πολιτική η οποία έχει μείνει αναλύωτη για 25 χρόνια. Πρέπει να απλοποιήσουμε λοιπόν τους κανόνες της προς όφελος των πολιτών μας και η κυρία Τόμας το είπε. Εγώ ενοχλούμε όταν βλέπω τους νέους να απαραίτούνται από την διεκδίκηση των κονδυλίων αυτών γιατί είναι πολύ χρονοβόρες και επαχθείς οι διαδικασίες. Η πολιτική μας όμως θα πρέπει να παραμείνει όπως είναι θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η πιο ορατή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών μας. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι η μόνη πολιτική η οποία έχει αυτή την άμεση επαφή με τους περιφερειάρχες, με τους δημάρχους, τους κοινοτάρχες, τους απλούς πολίτες. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει εκ μέρους της Κομισιόν, ώστε αυτή η πολιτική να μπορέσει να διατηρηθεί. Περιμένουμε τα πορίσματα αυτής της συζήτησης. Ούτως ή άλλως όμως είναι πολύ απαραίτητο η πολιτική συνοχής <clears throat> να απλοποιηθεί περισσότερο. Και όλα αυτά τα θέματα θα αντιμετωπιστούν στην μεταρρύθμιση των διαφορετικών πόρων και στην έκθεση για το Omnibus αλλά δεν μπορούμε να προσβλέπουμε σε σημαντικές αλλαγές μέσα στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Θέλουμε να δούμε τι μπορεί να αλλάξει χωρίς να δημιουργηθούν ε, ανασ... Ε, χωρίς να υπάρξει ανασφάλεια δικαίου σε σχέση με τους φορείς που εφαρμόζουν αυτή την πολιτική. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τις τωρινέ διαδικασίε, αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και περνάει από το χέρι μα για να ευνοήσουμε την εφαρμογή και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Μετά όμως από το 2020 θα ξεπεράσουμε την τωρινή κατάσταση. Έχουμε αρχίσει τη συζήτηση, αλλά υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για όλα τα διαφορετικά ταμεία. Δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλεκόμαστε σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εδώ έχουμε το μεγαλύτερο βάρος που υφίστανται οι αρχές στη διαχείριση των ταμείων γιατί είναι τόσο πολύ οι κανόνες, ενώ το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων έχει τόσο απλούς κανόνες, δεν πρέπει εμείς να έχουμε τόσο βαρύς και επαχθείς κανόνες. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα κοινό σύνολο κανόνων για όλα τα ταμεία με ελαφρές διαφοροποίησεις. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει αυτή η συζήτηση στην Κομισιόν, στο Κοινοβούλιο, επί το οποίο ποια είναι η άποψη των πολιτών και των εμπλεκομένων. Για τη σχέση των περιφερειακών Περιφερειακού Ταμείου και του Ταμείου Στατηγικών Επενδύσεων δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ταμείων, απλώς θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε καλύτερα τις δύο αυτές ενέργειες στα δύο αυτά ταμεία. Θέλουμε να έχουμε κάποια πρότυπα προγράμματα που δείχνουν πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και το Ταμείο Επενδύσεων δεν έχει γεωγραφική απλώ απλώς κάποια κράτη-μέλη είναι πιο έτοιμα να χρησιμοποιήσουν αυτό το ταμείο από άλλα. Πολλέ χώρε δεν έχουν τράπεζε οι οποίε είναι έτοιμε να αναλάβουν τον κίνδυνο χρήση του στρατηγικού ταμείου επενδύσεων. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με εμπειρογνώμονε. με... Μπορούμε να δίνουμε συμβουλέ στα κράτη-μέλη κατόπιν αιτήματο αυτών. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Έχουμε τόσα πολλά εργαλεία για να βοηθήσουμε και δεν λαμβάνουμε αιτήματα από τα κράτη-μέλη. Έχουμε 24.000 ανθρώπους επιτόπου στα 28 κράτη-μέλη και είμαστε έτοιμοι να στείλουμε ανταλλαγή απόψεων. Ε, να, δώσουμε, να ανταλλάξουμε ευέλτιστες πρακτικές. Αλλά δεν λαμβάνουμε αιτήματα από περιφέρειες, από κράτη-μέλη για ενημέρωση και βοήθεια να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυρία Τόμασιτς. Συμφωνώ μαζί σας κυρία Τόμασιτς ότι η απλούστευση είναι σημαντικότατη και όπως προανέφερα προσπαθήσαμε να το πετύχουμε αυτό μέσω της προτάσεως Omnibus. Περιμένουμε από το Ευρωκοινοβούλιο να ψηφίσει την πρότασή μας και ελπίζω ότι θα έχουμε άμεσο αντίκτυπο για τις ζωές των ανθρώπων διότι έχουμε καταρχάς ε, πρόταση για απλούστευση υπολογισμού του κόστους για την ε, συνοχή. Δεν χρειάζεται να μπαίνουν όλε οι αποδείξει ηλεκτρισμό για οποιοδήποτε, για κάθε έξοδο. Θα υπολογίσετε γενικό κόστος και βέβαια θα προχωρήσουμε και παραπάνω στην απλούστευση την περίοδο μετά το 2020. Αυτά μπορούσαμε να θεσπίσουμε σε αυτή τη φάση όμως. Ε, κύριε Γιακόβιτ, αναφερθήκατε στην αλληλεγγύη. Ε, δεν αποτελεί μυστικό ότι αυτή η πολιτική δέχεται πολλές ε, επιθέσεις. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό, διότι έχουμε τόσα πολλά προβλήματα. Δεν κατηγορώ κανέναν. Απλώς, ε, όπως σας είπα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες προκλήσεις, προβλήματα, μετανάστευση, το Brexit, δυσκολίες. Εσωτερική, εξωτερική ασφάλεια, Οπότε πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να πολεμήσουμε για τις περιφέρειες και τους Δήμους. Θέλουμε να ακουστεί η φωνή τους, διότι γνωρίζουν καλύτερα από εμά ε, τι πηγαίνει καλά, τι δεν πάει καλά και για πρώτη φορά ξέρετε κατά τη διάρκεια της προβληματικής περίοδου 2014-2020 τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον 5% ε, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που θα γίνεται διαχείριση των χρημάτων άμεσα από τους Δήμους. Από τις χώρες που γνωρίζω καλύτερα έδιναν 20% του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 35 πόλεις. Νομίζω ότι είναι μεγάλη ευθύνη αυτό Επίσης ε, είναι ένα σημείο εμπιστοσύνη αυτό ε, να έχουμε έργα και προγράμματα που πραγματικά τα αποκρίνουν τις ανάγκες του λαού. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι περιφέρειες και οι δήμοι θα έχουν ε, τη σύνοδο των Ευρωπαϊκών Πόλων, Eurocities, τον επόμενο μήνα. Θα έχουμε το φόρουμ για τις πόλεις Ξέρετε, συναντώμε με τις εκπροσώπους των πρωτεύουσών. Όταν μιλάμε για τις και για τις αστικές περιοχές, μιλάμε και συζητούμε και με εκπροσώπους των μεσαίων και μικρών πόλεων. Ο κύριος Φιλ Χόγκαν θα πρέπει να επανέλθει με κάποιες προτάσεις, διότι και μικρές πόλεις αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα παρόμοια με τις υπαίθρου. Πρέπει να συνεργαστούμε και κατά την άποψή μας αυτά τα, αυτοί οι πόροι για την υπαίθρο θα πρέπει να βοηθήσουν ούτω ώστε να αναπτυχθούν και τα χωριά της Ευρώπης. Κατά την άποψή μου, και είναι προσωπική άποψη αυτή, είναι επενδύουμε πολλά, παραδοσιακά πολλά χρήματα στις αστικά πυκνοκατοικημένες περιοχές και λησμονούμε την Ήπεθρο και διατρέχουμε τον κίνδυνο ε, να έχουμε πολύ ανεπτυγμένες πόλεις με ύπεθρο άδεια ε, και άδειε χώρες. Το συζητούσα αυτό με τον Φιλ Χόγκαν και είπα κατά την άποψή μου το Γερικό Ταμείο θα πρέπει να βοηθήσει και τα χωριά να αναπτυχθούν. Χρειάζεται συνεργασία για να κατασκευαστούν σχολεία, να πει το διαδίκτυο στην Ήπεθρο, θα βοηθήσει αυτό η οικονομική δραστηριότητα και να μην χρησιμοποιούνται μόνο για επιδοτήσει των γεωργών τα χρήματα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και όπως σας είπα νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και να εξασφαλίσουμε συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων και των διαφόρων τομέων. Τώρα για τις περιφέρειες, βέβαια η έποψή μου είναι ότι μέχρι τώρα δεν, πετύχαμε συνένεση για το ΑΕΠ ανακεφαλή. Υπάρχουν κάποιες ιδέες πώς πρέπει να ταξινομηθούν οι περιφέρειες διεξήχθη πολύ καλή συζήτηση στη Φλωρεντία με διάφορους ακαδημαϊκούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου και ο ΣΑ θα καταφτάσει με κάποιες ιδέες για δίκτυ ευημερία. Ε, συνδυασμός είναι αυτός, συνδυασμός μεταξύ ΑΕΠ ανακεφαλή ε, μαζί με άλλους δείκτες. Νομίζω πρέπει να είμαστε πραγματιστές όμως. Κατά άποψή μου το ΑΕΠ ε, κατακεφαλή ε, είναι κάτι ε, τυχαίο επίπεδο χαράς, ευημερίας κλπ. Πώς να βάλουμε τέτοιο δείκτη. Διότι μπορεί κανείς να είναι πανφτωχός ε, και να ε, είναι ευτυχισμένος, όπως στην Κούβα. Το ΑΕΠ κατά κεφαλή και η ποιότητα ζωής θα πρέπει να παραμείνουν οι βασικοί δείκτες. αλλά εγώ είμαι ανοιχτή. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Μπορούμε να δούμε το πώς θα εξετάσουμε το θέμα των περιφερειών. Με τις μειονεκτούσες περιφέρειες, βατικές περιφέρειες, πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, με βάση το ΑΕΠ κατά κεφαλή θα τις χωρίζουμε έτσι ή θα βάλουμε κάποια άλλα κριτήρια πολύ πιο ρεαλιστικά, όπως αεροκατοικημένες περιοχές, όπως η στέρηση. Τέτοια στοιχεία περισσότερο από τις δείκτης ε, ευημερίας. Ο κ. Παπαδημούλης. Με συγχωρείτε για την προφορά του όνοματό, σας. Λέει κύριε Επίτροπος, ξέρω ότι έχετε στεναρή θέση στον αφορά τη πολιτικής συνοχής και σας λέω ευχαριστώ γι' αυτό. Ε, γνωρίζετε πολύ καλά, ίσως καλύτερα από μένα, ότι δεν είναι πάντα σημαντικό το ποσό των πόρων, αλλά και το διοικητικό δυναμικό. Σχετικά με αυτό γνωρίζετε πολύ καλά ότι συνεργαζόμαστε στενά με τις ελληνικές αρχές για να αυξήσουμε το διοικητικό δυναμικό όσον αφορά την αλληλεγγύη. Εγώ μοιράζομαι, συμμερίζομαι την άποψή σας. Πρέπει να δείξουμε για την μετεγκατάσταση αυτή την αλληλεγγύη. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, αλλά προσφέρουμε τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τους πόρους μας. Δεν υποχρεώνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούμε μόνο το, τους πόρους για τη μετανάστευση και πράγματι η Ιταλία ζήτησε να αλλάξει η προγραμματική περίοδος. 2007-2013 για το Σικουρέτσα το πρόγραμμα να αγοράσει δύο σκάφη και βλέπετε κάθε εβδομάδα πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δύο σκάφη για τη διάσωση εκατοντάδων ζώων στη Νότια Ιταλία και η Ελλάδα έθεσε στο αποθεματικό κάποια, στην άβαλη, στην άκρη κάποια χρήματα για τη μετανάστευση. Η βοήθεια για τη μεταναστευτική κρίση δεν προήθε εις βάρος της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχής δεν πήρε κόπη επουδενή λόγω μεταναστευτικής κρίσης αλλά βέβαια θεωρώ ότι η πολιτική συνοχής μπορεί και θα πρέπει να βοηθήσει αν τα κράτη-μέλη ζητήσουν κάτι τέτοιο για την υποδοχή και ένταξη των ετούντων άσυλο. Κατόπιν αιτήματο του κράτους μέλους μπορούμε να κατασκευάσουμε νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, το κοινωνικό ταμείο μπορεί να συμβάλλει στην εκμάθηση γλωσσών, αλλά για τη μετεγκατάσταση. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με του εαυτού μα, διότι Φερρυπίν, η χώρα μου, είναι πρόθυμη να υποδεχθεί μετανάστε, αλλά δεν θέλουν να έρθουν. Και προσπαθούμε, και η Ρουμανία προσπαθεί να συμβάλλει με άλλου τρόπου, συμμετέχοντα στη Frontex ε, και σε άλλα μέσα. Ακόμα και στο Λουξεμβούργο δεν θέλουν να πάνε. Θα πρέπει να υπάρξει μια αλληλεγγύη που θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και βέβαια αν κάποια κράτη-μέλη όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα έχουν μεγαλύτερο βάρος να υπομισθούν, οι άλλοι θα πρέπει να βοηθήσουν και να δείξουν αλληλεγγύη. Πραγματικά ανησυχώ πάρα πολύ για αυτή τη διαίρεση, τη διαφορά που υπάρχει λόγω της μετανάστευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πάω στη Βαρσοβία με αυτό το μήνυμα, ότι θα πρέπει να δώσουν ένα μήνυμα αλληλεγγύης διότι δεν μπορούν να κατηγορούν συνεχώς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αφήνουν όλο το βάρος σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, μόνο και μόνο λόγω της γεωγραφικής θέσεως της Ελλάδας. Είναι πολύ σημαντικό να αποδειχθεί να εφαρμοστεί η αλληλεγγύη. Εν πάση περιπτώσει είμαστε έτοιμοι να επαναπρογραμματίσουμε την πραγματική περίοδο μας ζητηθεί. Άλλα κράτη-μέλη δεν χρειάζονται ένα προγραμματισμό. Είδα στη Γερμανία ε, τόσα πολλά υπέροχα έργα στο Βερολίνο στη Λιψία, στη Δρέσδη. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ακόμα και στα προάστια του Παρισιού είδα πολλά καλά πράγματα να γίνονται για τους μετανάστες. Ε, αυτό που θα πρέπει να αποφύγουμε είναι απομόνωση και διαχωρισμό, διότι αυτή η απομόνωση θα γίνει πυρηνική βόμβα για τις μελλοντικέ γενιές κατά την άποψή μου. Αυτή η γετοποίηση δεν πρέπει να συμβεί. Μία εβδομάδα πριν, κατόπιν ετήματος, αλλάξαμε το πρόγραμμα κατόπιν ετήματος των Βρυξελών, αλλάξαμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Βρυξελ, ε, και δώσαμε τα χρήματα στους γιατρούς του κόσμου. Έχουμε ένα κέντρο στο Μόλεμπεκ και στο Άντερλεχτ. Αλλάξαμε το πρόγραμμα κατόπιν ετήματος για να γίνουν κατάλληλες επενδύσεις για την φροντίδα των μεταναστών. Δώσουμε ευκαιρία. Τώρα, εκ των προτέρων αρισιμότητα θα σας δοθεί έκθεση πάνω σε αυτό τέλος ε, Μαρτίου. Όπως σας είπα, πέρα από το θέμα του ΑΕΠ θα δούμε και τι γίνεται με άλλα στατιστικά στοιχεία. Καλωσορίζω όλα σας τα σχόλια. Για μας όμως το ΑΕΠ παραμένει ένας βασικός ε, δείκτης. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο εκάλυψα ε, τα πάντα. Όπως σας είπα, κυρία Βάνα, ε, σκεφτόμαστε ενιαίους κανόνες για του, τα διάφορα ταμεία και οι εταιρικές σχέσεις σημαντικές, η κοινωνική διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική. Στο Omnibus έχουμε προτείνει να συνδυάσουμε τα διάφορα και το ΕΦΣΙ και το ΕΣΥΦ ε, και ελπίζουμε ότι αυτή η έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο και από το Συμβούλιο θα επιταχυνθεί ε, για να στηριχθεί η πρόταση Omnibus και να περάσει. Θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι υποφελή για τις επενδύσεις της περιφέρειας και ένας τέτοιος συνδυασμός πάντα θα αποφασίζεται από τις φορείς πολιτικής συνοχής και δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν. Τώρα, όσον αφορά την τεχνική προσαρμογή για την Ιταλία, η Ιταλία έλαβε 2,6 δις, έχετε δίκιο, είναι κυρίαρχη απόφαση των Ιταλικών αρχών το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ιταλία αυτά τα χρήματα αλλά συνομιλήσαμε με τον Υπουργό Ντεβιτσέντι και με εκπροσώπους των αρχών διότι γνωρίζουμε ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει με την μετανάστευση, την ανεργία. Επίσης ε, οι Ιταλικές αρχές αποφάσισαν να δώσουν 200 εκατομμύρια για τις τέσσερις ε, περιφέρειες. Ζητήσαμε να μας ενημερώσουν πώς θέλουν να μοιράσουν αυτό το ποσό και ξέρετε ότι υπήρξαμε αλληλέγγυοι, δώσαμε 30 εκατομμύρια ευρώ για το σεισμό, το, η, μέγιστη δόση μπορούσαμε να δώσουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης και τώρα περιμένουμε να γίνει αξιολόγηση των διαφόρων περιφερειών της Ιταλίας ώστε να γνωρίζουμε πόσα χρήματα πρέπει να καλύψουμε τι κόστος να καλύψουμε. Και υπήρξε μια πρόταση ότι πέρα από το Ταμείο Λιλεγγύης τα υπόλοιπα χρήματα ανακαλύπτονται 100% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη και περιμένουμε την απόφασή σας. Τώρα, όσον αφορά τη τεχνική προσαρμογή, είναι χρήματα που προέρχονται από το εξή, ότι η πραγματική κατάσταση διέφερε, ήταν χειρότερη από την πρόβλεψη. Οπότε σας αξίζουν αυτά τα χρήματα πέρα από το ποσό που σας δόθη. Δεν εναπόκειται σε εμά να αποφασίσουμε πώς θα πανώνται τα χρήματα. Εμείς απλώς προτείναμε να επενδυθούν αυτά τα χρήματα για την ενεργεία των νέων, τη μετανάστευση, διότι στην Ιταλία αποτελεί πρόβλημα και τώρα υπάρχει και το πρόβλημα λόγω των σεισμών. Ήταν απόφαση των Ιταλικών αρχών 200 εκατομμύρια να δοθούν στις τέσσερις περιοχές αυτές, αλλά μέχρι τώρα δεν λάβαμε λεπτομέρειες για το πώς θα μοιραστούν στις περιοχές τα χρήματα και για ποιους σκοπούς. Ευχαριστώ. Για το τελευταίο σχόλιο που κάνατε. Εγώ δεν ασκώ κριτική, δεν ξέρω, συγγνώμη κιόλας αν με παρεξηγήσατε, αλλά θέλω να πω ότι τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές τις αλλαγές. Οι πολίτες είναι πιο απαιτητικοί, ναι. Και πρέπει να μιλήσουμε για τα χρήματά μας, για τις επενδύσεις μας. Αν θέλετε μπορούμε να πάμε μαζί στην περιφέρειά σας και θα δείτε ότι μπορούμε να δείξουμε πολλές ε, περιπτώσεις που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι σίγουρη ότι όλοι γνωρίζουν ότι πολλές από τις θέσεις εργασίας που έχουν προέρχονται από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως ο κάθε πολιτικός παίζει τα χαρτιά του όπως νομίζει, αλλά η Ευρωπαϊκή Συνοχή δημιουργήθηκε για να καλύψει κενά. Τώρα γιορτάζουμε 60 χρόνια, την επέτειο 60 ετών τη συνθήκη τη Ρώμη. Σκεφτείτε πώ ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 60 χρόνια και σκεφτείτε πώ είναι τώρα. Είναι σαφές ότι για τα νέα κράτη-μέλη ήταν μεγάλη επιτυχία η διεύρυνση. Ε, μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη, αλλά 70 χρόνια επενδύσεων ανάπτυξης ειρήνης είναι κάτι μεγάλο, είναι το κοινό μας όραμα. Πρέπει λοιπόν να παλέψουμε για την Ευρώπη, για να παραμείνει ενωμένη, όπως είπε και ο κύριος Βανίστελ Ρόι. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καλύψουμε άλλα 7 ερωτήματα και τις απαντήσεις του στο επόμενο ένα λεπτό, οπότε να σας δείσω μία χάρη. Αν οι συνάδελφοι μπορούν να, σας, να μας στείλουν ε, γραπτός τις ερωτήσεις τους, να σας τις αποστείλουμε, να τις απαντήσετε αν μπορείτε. Και επίσης πρέπει να οργανώσουμε και μια έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσουμε την πολιτική συνοχή μετά το 2020 όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο να ακούσουμε τι διάφορε απόψει, να ακούσουμε τα ερωτήματα και να ακούσουμε βεβαίω και περισσότερες πληροφορίες από εσά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Καλή επιτυχία στην έκτακτη συνεδρίαση του Κολεγίου για τη Λευκή Βίβλο. Και περιμένουμε τις ερωτήσεις σας, συνάδελφοι, όσο δεν προλάβατε να πάρετε το λόγο, για να τις στείλουμε στην Επίτροπο. Ευχαριστώ για την κατανοησή σας, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο με την Επίτροπο. Συνεχίζουμε τώρα με το επόμενο σημείο της σήμερα της διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών. Το Συμβούλιο ιδρύθηκε το 1951 και είναι η συνολική οργάνωση ομπρέλα με 60 ε, ενώσεις μέλη από 21 χώρες ε, μιλώντας εξ ονόματος 150.000 ε, τοπικών ηγεσιών. Το Συμβούλιο προσπαθεί να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πολιτική ε, σε τομείς που έχουν ε, επιπτώσεις ε, στις, στους Δήμους και τις Περιφέρειες και παράσχει ένα φόρουμ συζήτησης μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών μέσω των εθνικών εκπροσώπων και των ενώσεών τους. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου ήδη τον Νοέμβριο του 2015 σήμερα. Θα κάνουμε άλλη μια ανταλλαγή απόψεων ε, για την δουλειά που κάνουν και για τη μελλοντική εργασία τους με την κυρία Καρόλα Γκιούνερσον, την ε, δήμαρχο της πόλης Σάλας στη Σουηδία, που είναι η εκπρόσωπος τύπου του Συμβουλίου για την πολιτική συνοχή. Οπότε συνεχίζουμε ουσιαστικά την ίδια συζήτηση που ξεκινήσαμε για την πολιτική συνοχή. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκίνερσον και μετά θα ακούσουμε τις απόψεις των μελών α, της Επιτροπής Ρέτζι, καταρχάς με τους συντονιστές. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Madam President. Πολύ σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε και η Πρόεδρος, είμαι Καρλα Γκούναρσον και είμαι δήμαρχος της Σάολαν που είναι ένας δήμος στην Σουηδία και επίσης είμαι ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Και έχω κρατήσει αυτή τη θέση για πολλά χρόνια. Με μεγάλη χαρά είμαι εδώ για την ανταλλαγή απόψεων μαζί σας για τα θέματα της πολιτικής συνοχής και ιδιαίτερα για τα τρέχοντα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί αλλά και για το μέλλον όταν ακόμα δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών είναι ένας ε, οργανισμός ομπρέλα των τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων και συναθρίζει εθνικές και περιφερειακές ενώσεις και μέσω αυτών εκπροσωπεί όλα τα επίπεδα των περιφερειών και δήμων στην Ευρώπη. Επομένως καλύπτουμε και το περιφερειακό αλλά και το τοπικό επίπεδο. Σήμερα <clears throat> περνάει μια δοκιμασία η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής. Μετανάστευση, χαμηλή ανάπτυξη, Brexit, που ήταν κυρίως η απόφαση περιφερειών που υπολείπονται οικονομικά και επίσης η και της άνοδου, της ανόδου λαϊκιστικών κομμάτων, όλα αυτά επισκιάζουν την μελλοντική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτουν να αμφιβόλο την προσθέμενη αξία που φέρνει στους πολίτες της Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καιρούς λοιπόν αβεβαιότητος, η δέσμευση για να εξασφαλίσουμε εδαφική συνοχή και ισορροπία και για να υπάρχει μια πολιτική συνοχή η οποία έχει νόημα για όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Και θέλω να υπογραμμίσω αυτά που είπε και η κυρία Επίτροπος για τη σημασία της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχής είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αντιληφθούν την ευρωπαϊκή πολιτική οι πολίτες. Έχει να κάνει με τα, τους ε, φορείς, τους δημοτικούς, με τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, με τις τοπικές αρχές που δίνει τη δυνατότητα λοιπόν αυτή η πολιτική σε όλους αυτούς τους φορείς να προχωρήσουν από κοινού μαζί. Είναι ένα εργαλείο για να καταδείξουμε στους πολίτες ότι η Ευρώπη νοιάζεται για αυτούς και είναι και ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κοινέ προκλήσεις με συντονισμένο τρόπο. Συμφωνούμε για όλες αυτές τις βασικές αρχές, αλλά συγχρόνω βλέπουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο αυτή η πολιτική έχει διατυπωθεί σήμερα μπορεί να μην είναι κατά αναγκή ο καλύτερος τρόπος για αύριο. Η μελλοντική πολιτική συνοχής θα πρέπει να καταδείξει ότι είναι το κατάλληλο εργαλείο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σε καθημερινή ζωή στους Δήμους και τις κοινότητές τους οι απλοί άνθρωποι. Το Συμβούλιο μας, το CMR, έχει αρχίσει τον προβληματισμό για το πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι κέρδε πολιτικές συνοχής μπορούν να εξακολουθήσουν να δίνουν σημαντικά ωφέλη με αποτελεσματικό τρόπο στους πολίτες μας, με ιδιαίτερη εστίαση στις περιοχές που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Στόχος μας είναι να υπογραμμίσουμε τους επόμενους μήνες τις κέρυες συστάσεις από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που ζητούν να υπάρξει μια μεταρρυθμισμένη πολιτική συνοχής πέραν του 2020. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου για πέντε σημεία εξονόματος αυτών που βρισκόνται στην πρωτοπορία της διαχείρισης και της μεταφοράς των ωφελών των ωφελών της πολιτικής συνοχής στους απλούς πολίτες κάθε μέρα, δηλαδή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Πρώτα απ' όλα, <clears throat> πιστεύουμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα στρατηγική για το επέκεινα του 2020 και αυτή η νέα στρατηγική θα έπρεπε να βασίζεται στους στόχους που ήδη έχουν τεθεί και θεσπιστεί για το 2030 σε ορισμένε πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης στις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα η βιώσιμη ανάπτυξη, η στοχή της βιώσιμης ανάπτυξης, Η στοχή της, κλιματικής, της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής των Παρισίων, του χάρη. Αυτές οι συμφωνίες πρέπει να δώσουν κατεύθυνση στην πολιτική συνοχή και να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξει πρόοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Επίσης θα πρέπει να διατηρηθεί και να διαβλεχθεί το πνεύμα της ενότητας και της αλληλεγγύης ό,τι αφορά την επίτευξη κοινών στόχων. Δεύτερον, η μελλοντική πολιτική συνοχή θα πρέπει να είναι περιεκτική. Δηλαδή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα εδάφη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς να λησμονεί αυτούς που βρίσκονται σε δύσκολες και κρίσιμες καταστάσεις, αυτούς που δεν έχουν υποδομές, τις περιοχές που έχουν λιγότερη καινοτομία, αυτές όπου υπάρχει ε, μεγάλος νέος πληθυσμός στις περιοχές που δεν φαίνεται να είναι ελκυστικές για το ιδιωτικό κεφάλαιο. Πρέπει κάτωθεν να λειτουργήσουν όλα αυτά βασιζόμενοι στην τοπική εμπειρογνωμοσύνη, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών των περιοχών και την οικονομική τους κατάσταση, για να δημιουργηθούν ελκυστικοί δημόσιοι χώροι και ευκαιρίες για όλους. Πρέπει επίσης να υπάρχει μια πολιτική η οποία έχει νόημα για όλους τους εμπλεκομένους εταίρους. Αυτή τη στιγμή η αρχή της εταιρικότητας δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως παντού. Ιδίως σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό των συμφωνιών εταιρικού χαρακτήρα και τα λειτουργικά προγράμματα, όπως καταδεικνύει και η μελέτη μας. Οι συναντήσεις συντονισμού δεν λαμβάνουν χώρα σε τακτά διαστήματα πάντα, ενώ μια πραγματικά αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής συνοχής απαιτεί οι διάφοροι κυβερνητικοί και φορείς αυτοδίκησης να λειτουργούν από κοινού. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η πολιτική να είναι πιο κοντά στους φορείς τοπικών αρχών, στις τοπικές αρχές και πιο προσβάσιμη σε αυτές. Να μπορέσει λοιπόν να υπάρξει μια καλύτερη εταιρική σχέση μεταξύ κεντρική εξουσία και τοπικών και περιφερειακών αργών. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα τη περίοδου προγραμματισμού, την εφαρμογή, την ε, υλοποίηση αλλά και τη φάση αξιολόγηση και παρακολούθηση τη πολιτική. Η μελλοντική πολιτική συνοχή θα πρέπει να εμπλέκει το τοπικό επίπεδο σε μεγαλύτερο βαθμό από στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, όχι μόνο στην επιλογή των προγραμμάτων και των σχεδίων, αλλά πάνω απ' όλα για την επιλογή των επενδυτικών προτεραιοτήτων σε κάθε περιοχή. Τα στοιχεία αυτά που υπάρχουν στον τωρινό κώδικα δεοντολογίας για την σχέση εταιρικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι δεσμευτικό ε, χαρακτηριστικό του μελλοντικού κανονισμού και όχι ένα χωριστό στοιχείο, κάτι το οποίο θα γεννήσει χωρίς αμφιβολία και διαφυσβητήσεις για το νομικό χαρακτήρα της, ένωσης, της έννοιας αυτής. Πρέπει επίσης να έχουμε μια ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη και μια στοχευμένη κατεύθυνση. Θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πολυεπίπεδες και πολυτομιακές στρατηγικές που να βασίζονται σε υποπεριφερειακούς προϋπολογισμούς και που θα επιτρέψουν μια καλύτερη συμμετοχή των τοπικών αρχών και των τοπικών εμπλεκομένων. Χρειαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ειδικά εργαλεία ώστε να μπορέσουμε να αποκεντρώσουμε στο βαθμό του δυνατού τις αποφάσεις. Το να έχουμε τοπικές επενδύσεις και ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο που τροφοδοτείται από την τοπική κοινωνία είναι σημαντικά για την επίτευξη των στόχων αυτών. Έχουμε δείξει στην έκθεσή μας ότι η απορρόφηση πολλές φορές περιορίζεται. Πολλές φορές θα πρέπει να υπάρξει και υποχρέωση των τοπικών αρχών να δίνουν τη δυνατότητα σε τοπικές και περιφερειακές αρχές ανεξάρτητα από το είδος τους να συμμετέχουν στα θέματα αυτά ακόμα και εάν οι διαχειριστικές αρχές θεωρούν ότι αναλαμβάνουν υπερβολική ευθύνη όταν αποκεντρώνουν τη λήψη αποφάσεων. Επίσης θεωρούμε ότι μια τέτοια προσέγγιση με πολλαπλά ταμεία είναι πολλές φορές δύσκολη στην εφαρμογή. Διότι υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες και διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τα διάφορα ταμεία. Γι' αυτό ίσως θα πρέπει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς ενιαίο κανόνα, ενιαίους κανόνες για τα πέντε ταμεία, να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ασφάλεια δικαίου ότι το τρόπος με μοναδική διαδικασία υποβολή αιτήσεων για διαχείριση και υποβολή αναφορών όσον αφορά όλα τα ταμεία. Τέταρτον, η πολιτική συνοχή θα πρέπει να απλουστευθεί ούτω ώστε να ενθαρρυνθεί η τοπική αυτοδίκηση για την πλήρη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων και με καλύτερο τρόπο από ό,τι κατά την τρέχουσα περίοδο θα πρέπει να είναι κάτι απλό, ευανάγνωστο και να κινητοποιεί διάφορες πολιτικές για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θα πρέπει να είναι πολύ περίπλοκη διαδικασία όσον αφορά τη δίκηση και τον έλεγχο. Φερρυπίν, σύμφωνα με την αξιολόγηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χάρη στην κυκλική οικονομία, 443 εκατομμύρια τόνοι αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσε να αποφευθεί και 180.000 άμεσες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μέχρι το 2030. Η τοπική αυτοδίκηση ε, στηρίζει αυτή την προσέγγιση. Γιατί όχι άλλωστε. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι χρειάζεται πρόσβαση στους αναγκαίους πόρους ούτως ώστε η φιλοδοξία να καταστεί πραγματικότητα. Πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πρόθυμη να έχει πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους. Όμως πόλεις με μικρότερες δυνατότητες πολύ συχνά αντιμετωπίζουν πάρα πολλά εμπόδια για την πρόσβασή τους στους πόρους. Απλούστευση λοιπόν και μείωση της γραφειοκρατίας είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Διαφοροποίηση όσον αφορά τους ελέγχους για τα κράτη-μέλη εκείνα που δείχνουν πολύ στεναρά εσωτερικά συστήματα είναι κάτι που συζητούν τα μέλη μας για το μέλλον. Τέλος, υπάρχει μια ανάγκη για θεσμικό δυναμικό, δημιουργία θεσμικού δυναμικού σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη και καλύτερη χρήση των θεματικών στόχων που ε, αφορούν την τεχνική αρρωγή δεν θα πρέπει να είναι κάτι που αφορά μόνο τις εθνικές αρχές αλλά και τους δικαιούχους. Θα ήταν χρήσιμο αυτό όσον αφορά τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κρατικών προμηθειών και χρηματοπιστωτικών μέσων. Αυτά κυρία Πρόεδρε είναι απλώς μία γεύση ε, των θεμάτων επί των οποίων σταζόμεθα. Αυτές οι συζητήσεις θα διεξαχθούν στην εκδήλωση ε, στις 28 Μαρτίου στις Βρυξέλλες του φορέα μας. Είσαστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε και να συμμετάσχετε στις συζητήσεις για το πώς θα διαμορφώσουμε το μέλλον της πολιτικής αυτής που είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο τώρα από ποτέ. Ο φορέα μας είναι πλήρω ε, αφοσιωμένο στη συνεργασία του με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκή Ένωσης για να προχωρήσουμε μαζί σε μια νέα πολιτική συνοχής μετά το 2020. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Συνάδελφοι, έχετε το λόγο. Αν έχετε ερωτήσεις, μην τυχόν έχετε κάποια σχόλια. Η κυρία Κρέου έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να μιλήσω πολύ καλά σήμερα. Γι' αυτό θα είμαι σύντομη. Υπογραμμίζω ότι όντω χρειαζόμαστε νέα στρατηγική για την μελλοντική πολιτική συνοχή. Νομίζω ότι του επόμενου μήνε θα πρέπει εντατικά να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση ενεργεία και την αντιμετώπιση τη ένδυα, Επιγόντως χρειαζόμαστε μια προτεραιότητα η οποία θα ασχοληθεί και στα πλαίσια της ψηφιακής, του ψηφιακού θεματολογίου για την για το συνδέεται άμεσα, άρρηκτα με την πολιτική συνοχή, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να θέσουμε μία προτεραιότητα ως προς το μέλλον, ως προς το όρομα που έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνώ μαζί σας ότι αυτή η αρχή της εταιρική σχέσης δεν θα πρέπει να μείνει θεωρία, θα πρέπει όντως να γίνει και πράξη και ίσως θα πρέπει να βρούμε νέους δρόμους που αυτό θα μπορεί να γίνει και πρακτικά και υποχρεωτικά ίσως. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει περαιτέρω κόστος διοικητικό και τα λοιπά για τα διάφορα project στο μέλλον. Αλλά έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Τους τελευταίους μήνες, τελευταίες εβδομάδες μιλάμε συνέχεια για περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη επικοινωνία, εσείς ως δήμαρχος πώς το βλέπετε αυτό. Οι πολίτες σας στην πόλη σας ξέρουν τι γίνεται μέσω, της, ε, των Ευρωπαϊκών Διορθωτικών Ταμείων στην πόλη σας. Υποθέτω ότι θα μπορούσατε και εσείς να τα κάνετε ό,τι κάνετε ακόμα καλύτερα. Πώς φαντάζεστε ότι μπορεί να βελτιωθεί η επικοινωνία και εμεί ω νομοθέτε εδώ μπορούμε να υποστηρίξουμε τι δικέ τις σα προσπάθειε, αλλά εσεί τι προτάσει έχετε να μα κάνετε, γιατί αυτό πραγματικά μα ενδιαφέρει ιδιαίτερω. Μιλάμε για δισεκατομμύρια και κανένα δεν ξέρει τελικά που καταλήγουν και σε τι μεταφράζονται. Θυμάμαι μια συνέντευξη κάποιον που τον ρώτησαν για ένα ευρωπαϊκό ε, project ε, που είναι, έχει, υπάρχει μια μεγάλη ταμπέλα που λέει συγχρηματοδοτούμενο project από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένας άνθρωπος που στέκεται μπροστά του και τον ρωτάνε τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πόλη σας και ενώ είναι μπροστά στην ταμπέλα δεν ε, λέει δεν ξέρω τίποτα. Πρέπει λοιπόν να μας πείτε κι εσείς πώς μπορούμε από τη θεωρία όντω να περάσουμε στην πράξη με συγκεκριμένε προτάσεις αν έχετε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ η κυρία Βάνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την κυρία Γκούναστον για τις ε, παρεμβάσεις, την παρέμβαση. Με ενδιέφερε ιδιαίτερα αυτό το οποίο αναφέρεται στο έγγραφο για το μέλλον της Ευρώπης. Για συντομία θα σας ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ερώτημα το οποίο ανέφερε και η κυρία Κρέλ για την αρχή της εταιρικότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ πέρα εμείς θέλουμε να τονίσουμε την ανάγκη ενίσχυσης και δεσμευτικότητα στην αρχή της εταιρικότητας. Μήπω μπορείτε να μας δώσετε όμω από τη δική σα εμπειρία και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα για την εφαρμογή τη αρχή τη εταιρικότητας από την έκθεσή τη και ένα άλλο θέμα που δεν έχει να κάνει με το μέλλον τη πολιτική συνοχή, αλλά για την δυνατότητα δράσης των, περιφερεια... των περιφερειακών, των ομοσπονδων κρατών και των δήμων Ποια είναι η αποψή σα σε σχέση με τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, παραδείγματος χάρη, για την συμφωνία ΤΙΖΑ που έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσιών. Εδώ υπάρχει πολύ σημαντικό περιθώριο για τη δράση των ομοσπόνδων κρατών και φυσικά υπάρχει μια σειρά ρήτρα, ρητρών για την κοινοτικοποίηση ορισμένων υπηρεσιών και εδώ φυσικά υπάρχει το ερώτημα του ποιος έχει το δικαίωμα να ασκεί την ρυθμιστική εξουσία σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών. Θα με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σας. Ευχαριστώ. Άλλα ερωτήματα. Δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα. Να κάνω και εγώ ένα ερώτημα, λέει η πρόεδρος. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ. Ο στόχος μας σήμερα αυτός είναι στην Επιτροπή Ρέτζη να ακούσουμε την φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας στην συνεδρίασή μας και για τη συνέχιση της εταιρική μας σχέσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε τις πληροφορίες που αναφέρετε και να σας εμπλέξουμε στην συζήτησή μας. Λόγω της αρχής της λόγω της ανάγκης να υπάρχει ορατότητα της πολιτικής συνοχής Λόγω όλων αυτών των θεμάτων και των προβλημάτων που είναι αντικείμενο συζήτηση εδώ, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω να μας πείτε ποια είναι και τα δικά σας οράματα. Αν βλέπετε στο μέλλον της πολιτικής συνοχής, όπως είπε κάποιος συνάδελφός μου, να υπάρχει μια ομαλή μετεξέλιξη της τωρινής πολιτικής ή αν βλέπετε μια επανάσταση η οποία εκ βάθρων θα αλλάξει τη μορφή αυτής της πολιτικής. Χρειαζόμαστε λοιπόν σταθερότητα και ένα μακρύ ορίζοντα που θα μας δώσει τη δυνατότητα να βλέπουμε μακροχρόνια αποτελέσματα ή θέλουμε ραγδαίες αλλαγές. Ποια είναι η δική σας άποψη λοιπόν μεταξύ των μελών σας, ποιες απόψεις επικρατούν. Ευχαριστώ. Έχετε λοιπόν τα ερωτήματά μας. Απαντήστε λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ας ξεκινήσουμε από το τοπικό επίπεδο. Το ερώτημα ήταν αν εμείς καταφέρνουμε να κάνουμε τους πολίτες να συμμετάσχουν και να γνωρίζουν οι πολίτες μας ποια είναι τα διάφορα προγράμματα που έχουμε στο Δήμο μας ή στην γειτονιά μας. Την ευρύτερη. Καταρχάς να πω ότι βέβαια εγώ και οι συνάδελφοί μου μπορούμε να είμαστε πολύ καλύτεροι Ταυτόχρονα όμως θα ήθελα να πω ότι καταρχάς χρειαζόμαστε περισσότερο δυναμικό πρέπει να δημιουργηθεί. Όταν μιλάμε για δυνατότητες, ικανότητες και δυναμικό και δημιουργία αυτού θα πρέπει να εμπλακεί στην προσπάθεια κοινωνία των πολιτών. Όχι μόνο οι διαχειριστικές αρχές σε εθνικό επίπεδο, διότι αν ο κόσμος έχει περισσότερες πληροφορίες, τότε θα θέλει να συμμετέχει και περισσότερο στις όλες τις προσπάθειες και τα έργα. Νομίζω ότι όταν διεξάγονται συζητήσεις σε τοπικό επίπεδο περί επικειμένων έργων και προγραμμάτων προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο να συμμετέχει στις συζητήσεις. Ακόμα και αν δεν γνωρίζουμε αν στο τέλος θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα ή όχι. Προσπαθούμε όμως ε, να διεξαγάγουμε τη συζήτηση με κοσόπους κοινωνίας των πολιτών, με τους πολίτες, για να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συζητήσουν και να συμμετέχουν στις συζητήσεις. Διότι δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση αν καθόμαστε στο Δημαρχείο. Αν καθίσω εγώ στο Δημαρχείο, στο Δήμο μου και αποφασίσω ότι να αυτό θα είναι το έργο για το Δήμο μου, τότε δεν μπορώ να πετύχω, αλλά μπορούμε να πετύχουμε εάν έχουμε συμμετοχή του κόσμου, σε ευρύ φάσμα, ευθύ εξ αρχής να συμμετέχει ο κόσμος και βέβαια κάτι απλούστατο. Ίσως να γελάσετε, αλλά θα σας πω ότι το σημαντικότερο είναι να διαδίδεται η γνώση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ωφέλη που αποκομίζει κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι να προβάλλουμε τη σημαία με τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όπου υπάρχουν έργα και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όπου υπάρχουν δραστηριότητε χρησιμοποιούμε αυτή τη σημαία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι για κάποιου αυτή είναι η μόνη διασύνδεση που μπορούν να δουν και να καταλάβουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν βλέπουν το σημαίακι ε, θα πρέπει να λησμονήσουμε ε, τη συζήτηση για το μέγεθος, θεωρητικέ θεωρητικές συζητήσεις, να δούμε πώ μπορούμε να συμβάλλουμε εμεί στο έργο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας. Αυτό είναι το βασικό θέμα συζήτηση. Αλλά πάντα θα πρέπει να λέμε ότι αυτό είναι ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το ρόλο παίζει. Στο Δημαρχείο μου πάντα χρησιμοποιούμε την Ευρωπαϊκή Σημαία, παραδείγματο χάρη. Μαζί με τη Σουηδική Σημαία και τη Σημαία του Δήμου. Έχουμε και την Σημαία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορά που χρειάζεται να το δείξουμε αυτό στον κόσμο. Θα ήθελα να πω λοιπόν, θέλουμε συμμετοχή του λαού σε πολύ πρώιμο στάδιο. Δημιουργία δυνατοτήτων, δυναμικού, ούτως ώστε να μπορεί ο κόσμος να μπορεί να συμμετέχει στην όλη διαδικασία. Θέλουμε ορατότητα μέσω της χρήσης της σημαίας ή με άλλους τρόπους για να δείχνουμε ότι αυτό που γίνεται γίνεται χάρη σε βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα όταν συζητούμε το μέλλον, κατά πόσον πρόκειται περί επαναστάσεως ή περί σταθερότητας, καμιά φορά, ξέρετε, όταν χρειάζεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνει κάτι κανεις θεωρεί ότι είναι καλύτερη επανάσταση. Αλλά για να διευκολυνθούμε εμεί σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, εγώ θα επιθυμούσα να έχω σταθερότητα. Αλλά μια σταθερότητα ε, με πολλές αλλαγέ. Πρέπει όμως να υπάρχει και μια βάση γι' αυτό. Να μπορούμε να σταθούμε και να προχωρήσουμε εκεί πέρα. Διότι χρειάστηκε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να μάθουμε τι γίνεται με τα διαθωτικά ταμεία. Και ακόμα δεν καταλαβαίνουμε πώς να τα χειριστούμε. Εάν δεν τα μάθουμε αυτά, δεν αλλάξουμε πολλά θα πρέπει να ισχύουν όλοι οι κανόνες για όλα τα ταμεία. Αν γίνει αυτό, γίνουν τα πράγματα πολύ εύκολα. Έχουμε σταθερότητα, αλλά μπορούμε και να προχωρήσουμε και δημιουργούνται περισσότερες δυνατότητες για τον κόσμο να μπορεί να συμμετέχει στην όλη προσπάθεια και στο όλο έργο. Τώρα οι και οι διαγωνισμοί, οι κρατικές προμήθειες. Χρειάζεται μια ξεχωριστή συνεδρίαση για αυτό το θέμα, διότι σε τοπικό επίπεδο το θέμα αυτό των ε, φοδιασμών και προμηθειών του δημοσίου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα ούτως ώστε οι κρατικές προμήθειες να γίνονται με τον σωστό τρόπο ταυτόχρονα να μπορούμε να πετυχαίνουμε και τους στόχους του Δήμου διότι πάντα πρέπει κανείς όλα αυτά να τα συνδυάζει σαν ντόπια πολιτικός έχω στόχους. Αυτή είναι η στόχη μου, λέω. Και μετά το θέμα των διαγωνισμών και των κρατικών προμηθειών είναι ένας τρόπος για να πετύχουμε τους στόχους σε τοπικό επίπεδο. Αυτά. Ακάλυψα κάποιες από τις ερωτήσεις και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων με, την εκπρόσωπο του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών. Βεβαίως είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στις μελλοντικέ μας συζητήσει. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξη. Η συγγήτριά μας, η κυρία Κρέλ, θα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότηση για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο Γενικό Προπολογισμό της Ένωσης. Είναι η πρόταση Omnibus. Η Επιτροπή μας προετοιμάζει γνωμοδότηση για κάποια από τα άρθρα της ε, πρότασης αυτής, όπου έχουμε ε, αποκλειστική αρμοδιότητα. Και η κυρία Κρέλ θα μας, θα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής της. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Η πρόταση της Κομισιόν, η βασική της στοχοθέτηση είναι η απλούστευση των ε, δημοσιονομικών κανόνων και άρα και η απλούστευση της πολιτικής συνοχής. Αυτό το υποστηρίζουμε, το υποστηρίζω εγώ απολύτως και γι' αυτό στον τομέα αυτό υπάρχουν λίγες αλλαγές που θα ήθελα να κάνω από τη δική μου, μέσω της δικής μου γνωμοδότησης σε σχέση με το τι μπορεί να απλουστευθεί. Έχω ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την, τα απλουστευμένα κόστη και τις επιλογές που μπορεί να είναι υποχρεωτική η διάταξη όπως προτείνει η Κομισιόν. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε λίγο μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη, να τους δώσουμε περισσότερη ευελιξία και στις περιφέρειες και στα κράτη-μέλη. Γιατί μπορεί μετά από τρία χρόνια, ας πούμε, της εισαγωγής αυτών των νέων κανόνων, ε, να έχουν συνηθίσει όλοι να κάνουν ε, τους, ε, τους υπολογισμούς έτσι όπως πρέπει. Αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι αφού είναι τόσο δυσχερές αυτό το σύστημα δεν μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο απλό. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ η υποχρεωτική χρειά αυτής της διάταξης θα πρέπει να αφαιρεθεί από την πρόταση να μπορούν δηλαδή τα κράτη-μέλη να την ε, χρησιμοποιήσουν, αλλά να μην πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη διάταξη αυτή. Φαντάζομαι ότι θα, γίνει από, θα χρησιμοποιηθεί από πολλέ ε, περιφέρειες αυτό, αλλά αν είναι πολύ περίπλοκο, τότε θα πρέπει για να έχουμε τα ωφέλη που θα φέρει αυτή η απλούστευση να είναι εθελοντικό το σύστημα αυτό. Τώρα, οι αλλαγές που έκανα εγώ και που προτείνω στο έγγραφό μου επικεντρώνονται κυρίως εκεί που γίνεται παρέμβαση στην ε, πολιτική συνοχής. Μία πρόταση της ε, Κομισιόν με βρίσκει το σύμφωνη, η επιπλέον προτεραιότητα που εισήχθη στην έκθεση για το θέμα των προσφύγων και της μετανάστευσης. Να δοθεί λοιπόν στήριξη σε αυτό και το Ταμείο Συνοχής να, είναι, να χρησιμοποιηθεί για την υποδοχή και για την ένταξη των προσφύγων στα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι αυτό είναι απολύτως σκόπιμο, απολύτως λογικό και δείχνει ότι ακόμα και σε μια δύσκολη περίοδο μπορούμε να παρέμβουμε με ε, και να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες προκλήσεις. Και αυτό μπορεί να γίνει με αρκετά απλό τρόπο, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μην επιβαρυνθούν επιπλέον, ούτε οι περιφέρειους. Επίσης, προτείνω μία αλλαγή σε ό,τι αφορά τις ε, υποδομές ε, μικρής κλίμακος. Κυρίως ε, για τον τομέα του πολιτισμού. Εδώ η Κομισιόν προτείνει μια πλήρη απελευθέρωση του, του ύψους των κορδιλίων που μπορούν να διατεθούν εγώ προτείνω, έχοντας υπόψη ότι και στην τελευταία θητεία είχαμε παλέψει για να υπάρξει περιορισμός των κονδυλίων γιατί τα πολιτιστικά μνημεία είναι πραγματικά ένας πολύ σημαντικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν είναι στην ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γι' αυτό είχαμε περιορίσει τα ποσά σε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία αλλά βλέπω από τις ε, περιφέρειες να ζητείτε περισσότερη ευελιξία. Γι' αυτό προτείνω ο ορισμός, τι είναι δηλαδή μια μικρής κλίμακος υποδομή, να αλλάξει. Και προτείνω να πούμε ε, project μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ. Και για project που έχουν να κάνουν με πολιτιστική κληρονομιά, ε, να έχουμε ένα όριο 20 εκατομμύριων ευρώ και βεβαίως σε αιτιολογημένες ε, περιπτώσεις να μπορούν να δοθούν και υψηλότερα ποσά. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη έτσι από τη μία θα μπορούν να δείξουν περισσότερη ευελιξη και από την άλλη θα καταστεί σαφέ ότι εδώ δεν. Ε, δεν είναι μια πηγή που δίνει-δίνει χωρίς τελειωμό αλλά ότι υπάρχουν και κάποια όρια για αυτά τα project. Και νομίζω ότι για, το μέλλον, για τη συζήτηση που θα κάνουμε για το μέλλον τη πολιτική συνοχή, είναι σημαντικό αυτό, γιατί πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι και στο μέλλον θα πρέπει να επενδύσουμε και στους πολίτες μας και γι' αυτό δεν μπορούμε να, υπερβάλλω λίγο, αλλά δεν μπορούμε να επενδύουμε σε ξεχασμένες πέτρες συνέχεια. Αυτό λοιπόν μπορεί να αποτελέσει ένα κομμάτι της συζήτηση για τη μελλοντική πολιτική συνοχή. Τώρα, κάτι άλλο που προτείνω. Η σύνδεση των προγραμμάτων, των επενδυτικών του προγραμμάτων και της ε, πολιτικής συνοχής. Ξέρετε ότι ήδη υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει συνδυασμό εργαλείων, συνδυασμό μέσων. Υπάρχουν παραδείγματα για το πώ γίνεται αυτό. Η Κομισιόν ε, όμω προτείνει ένα μέσο το οποίο πάει επέκεινα των όσων συνέβαιναν μέχρι τώρα. Κάθε την δική μου άποψη, εδώ χρειαζόμαστε περισσότερη διαβούλευση. Προτείνεται ένα μέσο, νομίζω η κυρία Βάνα το είχε αναφέρει, Προτείνεται λοιπόν ένα μέσο, σε θελούσια βάση, ναι, αλλά χωρίς κανένα ανώτατο όριο. Διατίθενται χρήματα από το Ταμείο Συνοχής για το πνευματικό πλάνο του Γιούγκερ. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την πολιτική συνοχή, είναι τελείως άλλος ορισμός εκεί. Οπότε από την, ε, παίρνουμε λεφτά από την πολιτική συνοχή για λόγους διοικητικού και τα βάζουμε σε, άλλα, σε άλλες γραμμές του προπολογισμού και από την πρόταση Κομισιόν δεν ξεκαθαρίζεται το ότι αν ας πούμε η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Πολωνία βάλουν χρήματα στο, ε, διαθέσουν χρήματα, τα project θα χρηματοδοτηθούν και θα πρέπει να πάνε τα χρήματα πίσω στις χώρες οι οποίες τα έβαλαν στο συγκεκριμένο ταμείο. Χρειάζεται λοιπόν εδώ να υπάρξει έντονη συζήτηση. Ε, την κάναμε στην προηγούμενη θητεία όταν χρειάστηκαν 10 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για να, κάνουμε το, για να υποστηρίξουμε το Connecting Europe Facility το οποίο είναι πραγματικά μια πολύ σκόπιμη διαδικασία, αλλά βεβαίως τα κράτη-μέλη τα οποία τα έπληξε αυτή η, ε, αυτή η απόφαση α, ε, αναρωτήθηκαν εγώ θα πάρω τα χρήματα που έβαλα πίσω για τα δικά μου τα project. Και αυτό χρειάστηκε και κόστο και χρήμα και χρόνο και συζητήσει με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο και εδώ εντό του οίκου μα, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια πρόταση η οποία θα πηγαίνει προ τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, βεβαίω πρέπει να είναι δυνατή η παρέμβαση σε εδαφικό επίπεδο, αλλά μια τέτοια παρέμβαση δεν θα προβλέπεται για τα επενδυτικά προγράμματα. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και από κοινού με τη συζήτηση που θα κάνουμε για το μέλλον της πολιτικής συνοχή. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε αρπακόλα και αν δούμε και τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε και πρέπει να τα τηρήσουμε. Φυσικά ο τίτλος της έκθεσης λέει απλούστευση και η Επιτροπή μας Βεβαίω δεν είναι αντίθετη με τι ε, απλουστεύσει, ούτε θέλει να τι καθυστερήσει. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι κατα... πάρα πολύ σωστό ε, να έχουμε την ε, συζήτηση και, για το, για και στα πλαίσια του ΕΣΥΦ και του ΕΣΦΗ και να καταλήξουμε τελικά σε μια καλή συζήτηση έτσι ώστε η Κομισιόν να έχει μια καλύτερη πρόταση στο τραπέζι. χρειαζόμαστε χρόνο λοιπόν για να αναλύσουμε ποια είναι τα συμφέροντα της πολιτικής συνοχής και πώς μπορούμε να έχουμε έναν λογικό σύνδεσμο, μια λογική συνεργασία των δύο μέσων και τι μπορούμε να αλλάξουμε. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο μέσα έτσι ώστε να επιφέρουμε ανάπτυξη μέσω αυτών στα κράτη-μέλη. Η έκθεση της Νομίζω ότι δεν είναι απολύτω ε, ισόρροπη, αλλά δεν ε, είναι και πολύ μακριά από την ισορροπία, οπότε δεν έκανα δραστικέ αλλαγέ. Αρκεί όμω να γίνει αυτή η έξτρα συζήτηση που χρειαζόμαστε. Τώρα τα θέματα της νομοθεσίας για τα νέα α, τις νέες ρυθμίσεις για το επενδυτικό σχέδιο εμείς δεν έχουμε ακόμα απόλυτη γνώση. Το Κοινοβούλιο ακόμα συζητά για το πώς θα μπορέσει να συζητήσει για το μέλλον του επενδυτικού σχεδίου. Επομένως είναι κάπως πρόοδο να συνδέσουμε την πολιτική συνοχή με το σχέδιο στρατηγικών επενδύσεων. Ελπίζω όμως ότι παρόλα αυτά υπάρχει συνένεσή σας για αυτό το σχέδιο και θα μπορέσουμε με την Κομισιόν, με γαλήνη και με συζητήσεις να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αλλά χωριστά από τη διαδικασία του Omnibus. Πιστεύω λοιπόν ότι σε γενικές γραμμές είναι όλα αυτά που είχα να σας πω, μα ξέχασα κάτι ακόμα βέβαια. Η Κομισιόν για τη διαδικασία αυτή απλοποίησης είχε αναφέρει την έννοια της διαφοροποιημένης αντιμετώπισης των επενδυτών. Για μένα από την πρόταση αυτή της Κομισιόν όμως δεν προκύπτει για ποιους ακριβώς αναφέρεται. Είχα ζητήσει λοιπόν από την Κομισιόν να μας εξηγήσει καλύτερα, να μας δώσει ένα ορισμό, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα. Και από ό,τι βλέπω θα μπορούσαμε ίσως η Κομισιόν να μας δώσει ε, ένα τέτοιο ορισμό να περιλάβουμε στις αιτιολογικές σκέψεις, να, μπορούσουμε, να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια τροπολογία στην έκθεση, γιατί αλλιώς θα έχουμε κάποιες ε, δυσκολίες. Δεν θα ξέρει να σε παιδιτής αν υπόκειται σε αυτή την απλοποιημένη διαδικασία ή όχι. Και θα πρέπει να ξέρει λοιπόν με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν κατεπηγόντως αν μπορέσει να μας δώσει μια απάντηση σε σχέση με τη φύση αυτής της διαφοροποίησης και τον ορισμό ο οποίος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία με όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Τους ευχαριστώ ήδη. Προβλέπετε αυτή η εβδομάδα γίνει και μια συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές. Σας παρακαλώ όμως επιπλέον <clears throat> οι τροπολογίες που θα καταθέσετε και που ελπίζω θα λάβω υπόψη. Να μην έχουν σαν στόχο να αλλάξουν το σύνολο του, της νέας αυτής οδηγίας, αλλά να αλλάξουν ε, πλήρω τον κανονισμό μάλλον αυτών, αλλά να μπορέσουν να εστιάσουμε ακριβώ τα στοιχεία που έχει αναφέρει η Κομισιόν και ελπίζω και προσβλέπω συνεργασίας. συνεργασίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ανέφερα στην αρχή ότι έχουμε δύο επιλογές όσον αφορά τις τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα, τα μέλη μπορούν να προτείνουν τροπολογίες άμεσα στην Επιτροπή Ρέτζι για το χρησιμοποιητικό κανονισμό, το κομμάτι αυτό της προτάσεως και για τα άρθρα που αφορούν στις αποκλειστικές μας αρμοδιότητες αυτού του είδους οι τροπολογίες μπορούν να παραδοθούν στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα άρθρα της προτάσεως, για τα οποία άλλες επιτροπές έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα εκτός από τη Ρέτζη, σύμφωνα το άρθρο 54, Επιτροπή Επασχόλησης, Γεωργίας, ε, Τραν και Ήτρε, τα μέλη μας εκεί καλούνται να υποβάλουν τις τροπολογίες τους άμεσα στις αντίστοιχες αρμόδιες επιτροπές και αυτές θα τις συμπεριλάβουν στις εκθέσεις τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Να προτείνετε προθεσμίες τροπολογίες στην Επιτροπή μας 3 το απόγευμα στις 7 Μαρτίου, Τρίτη. Έχουμε μία εβδομάδα για τις ε, τροπολογίες. Τώρα, μετά από αυτές τις διευκρινήσεις, να δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές Ξεκινώντας από τον κύριο Βαν Νίστελροϊ, καταρχάς να σας συγχαρώ κυρία Πρόεδρε για την άριστη διαχείριση των απογευματινών μας εργασιών. Θεωρούσα ότι θα ξεκινούσαμε στις 5. Αλλά έχουμε κινηθεί πιο γρήγορα. Έχασα λοιπόν την παρουσίαση, την προφορική της συγγήτριας, για να είμαι ειλικρινής. Θα είμαι πολύ σύντομος. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως στη συζήτηση με την παρουσία της Επιτρόπου, θέλουμε να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε το ΕΦΣΙ σε σχέση με τους πόρους μας του ΕΖΙ και να δούμε τις λεπτομέρειες. Διότι πρόκειται περί διαφορετικών εργαλείων. Όπως είπε η Επίτροπος, δεν υπάρχει κάποιο γεωγραφικό κριτήριο που περιέχεται. Αν εξετάσουμε εν γέννη το εύση, τελικά θα έπρεπε να προβλέπονται γεωγραφικά κριτήρια. Δεν υπάρχει περιφέρεια, κυρίως της ΝΑΤΣ 2, που βάζει τα 10% των πόρων. Στη συνδυασμένη χρηματοδότηση μπορεί να μπει σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο αυτό το ποσό που παίρνει χρήματα από το ΕΦΣΙ και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ERDF. Εκ των προτέρων όμως θα πρέπει να είναι κανείς βέβαιος ότι αυτά τα προγράμματα καταλήγουν στην ε, περιοχή σου, αλλιώς δεν θα το ξεκινάς, δεν το κάνεις. Καλό και άγιο να λέει κανείς ότι μπορεί να φέρει χρήματα από το ERDF ε, για έργα που δεν ξέρει όμως κατά πόσο θα ε, όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, η μεγάλη συνεισφορά του Περιφερειακού Ταμείου, των Περιφερειακών Ταμείων, είναι ότι κινούνται οριζόντια, συντονισμένα. Αυτή είναι η προσέγγιση, όπως την περιέγραψε η Επίτροπο το απόγευμα. Πράγματι, μιλάμε για ανθρώπους, δημιουργία δυναμικού, για επιχειρήσεις, επιχειρηματικά θέματα, υποδομές, ε, όλα από κοινού. Άρα χρειάζεται μια καλή προετοιμασία μέσω θεματικής συγκέντρωσης και άλλων συναφών προσεγγίσεων. Θέλω να ξέρω περισσότερα. Και η κυρία Κρέλ θέλει να γνωρίζει περισσότερα. Και τίθεται το εξή ζήτημα. Πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε. Πώ μπορούμε να κρατήσουμε το σωστό πλαίσιο για τους πόρου ΕΣΥ, αλλά να μην αρνηθούμε ιδιωτικέ επενδύσει ή χρήματα του ΕΦΣΥ. που θα αποτελούν εγγύσει για κεφάλαια κινδύνου, τραπεζικέ επενδύσει, συνταξιωτικά ταμεία κλπ. Επενδύσει συνταξιωτικών ταμείων κλπ. σω μπορούμε να προτείνουμε κάτι μέσω τροπολογιών. Η εδαφική προσέγγιση να πλησιάσει περισσότερο την πραγματική ζωή. Έκανα το ίδιο εγώ, το θυμάμαι. Όταν ετοίμασα γνωμοδότηση. Ετοίμασαμε γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ. Και ήμουν εισηγητή και είπα να δούμε πώς λειτουργεί, είναι κάτι διαφορετικό. Να δούμε ποια θα είναι η εμπειρία μας, να δούμε αν πρέπει να αλλάξουμε τους ε, κανόνες. Αυτή ήταν η προσέγγιση μου τότε. Διότι εγώ υποστήριζα συνέργειες αν ε, εκτελούνται τα έργα αποσπασματικά, αυτό δεν επιτυγχάνει. Ίσως θα ήταν συνετό αύριο να συναντηθούμε και στη συνάντηση ίσως θα μπορούσατε να πείτε μέχρι 10-15% των πόρων του ΕΖΗ μπορούν να μπουν σε ένα διάνυμα, σε ένα φορέα για να προωθηθεί. Αυτό προβλέπετε τους κανονισμούς και το κάνετε και το εύση αυτό. Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να βρεθεί μια λύση. Να μην περιμένουμε μέχρι να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την επόμενη περίοδο. Κατά την άποψή μου, το ΕΦΣΙ θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί η κάλυψή του και θα ενισχυθεί το ΕΦΣΙ. Ίσως να ενταχθεί στο πλαίσιο είναι η καλύτερη λύση και να μπούμε σε αυτή την προσέγγιση. Πριν χάσουμε το τρένο. Γιατί το τρένο έφυγε. Άμα φύγει, έφυγε. Πάντα το τρένο. Έχουμε μοναδική ευκαιρία τώρα να αλλάξουμε τον κανονισμό. Και το δεύτερο που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα εγώ το ευχαριστήθηκα το απόγευμα διότι ο Επίτροπο μα είπε ότι θέλει να ετοιμάσει σχέδιο δράση όσον αφορά την επικοινωνία, την ορατότητα, κάπω έτσι το έθεσε. Και το υποσχέθηκε. Ήδη είδα κατά πόσο μπορούμε να έχουμε κάποια τροπολογία που θα υποβάλουμε, ούτω ώστε να επιφέρουμε κάποιε προσαρμογέ μικρέ. Φερρυπίν, όταν τελειώνει ένα έργο τώρα, όπω είπε ο Επίτροπο, καμιά φορά δεν φαίνονται τα ευρωπαϊκά άστα τη σημαία αυτό δεν είναι θέμα επικοινωνία. Απλώ δείχνουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν ευρωπαϊκή πόλη με αυτό το σημαίακι. Τι εννοώ εγώ. Τα διευθυντικά ταμεία να, να φαίνεται ότι δίνουν αποτελέσματα σε 4-5 χρόνια. Τότε θα πρέπει να εκφράζονται οι οποίοι ωφελούνται από τις επενδύσεις μας. Δεν αφορά μόνο τη στιγμή που ολοκληρώνεται το έργο, αλλά μετά. Αυτό αφορά την επικοινωνία. Εξέτασα κάποιες δυνατότητες να κάνουμε κάποιες αλλαγές, κάποιες τροπολογίες και συμφωνώ με κάποιο παράδοξο. Η πρώτη απάλεια, απώλεια, συγγνώμη, που, που έχει αναφερθεί συχνά από συναδέλφους, ότι πρέπει να ακολουθήσουμε σωστή προσέγγιση. Κατά λοιπά. Ας καθίσουμε, ας συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν δούμε μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος κοιόδης, ο κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υποστηρίζω τις προτάσεις που έκανε η συγγήτρια κυρία Κρέλ όσον αφορά την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των ενδιαφερομένων που θέλουν να επιλέξουν το αίσιο αλλά να μην επιβαρύνονται αυτοί που δεν είναι έτοιμοι να εγκρίνουν αυτή την προσέγγιση. Η Επιτροπή Ρέτζη θα πρέπει να δείξει κατανόηση για τις διάφορες δυνατότητες που υπάρχουν ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η απλούστευση σε ένα κάτω μέλος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρξει απλούστευση και σε άλλα κράτη-μέλη θα πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς, να είμαστε πιο διαφανείς όσον αφορά θέματα που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία μας. Στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων περί των διατάξεων Omnibus, η συγγήτρια κυρία Κρέλ είπε ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν συμφώνησε ακόμα το πώς αυτό θα πλουστεύσει τη διαδικασία και ποια είναι η πιο ενδεδειγμένη προσέγγιση όσον αφορά την επίτευξη της απλούστευσης άνευ ε, περιπλοκών στη διαδικασία και χωρίς να αυξάνεται το άχθος που βαρύνει τα κράτη-μέλη. Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτή η αναγκαία ευελιξία, η πρόταση εμπεριέχει διατάξεις περί αυξήσεως του ορίου και διατηρήσεως της υποδομής μικρής κλίμακας. Είμαι κατά αυτών, είμαι κατά των τροπολογιών 1, 8 και 9 διότι πιστεύω ότι αυτά τα ανώτατα όρια δεν θα οδηγήσουν σε απλούστευση, αλλά θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο για πολλά κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι στην πρότασή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει εισαγάγει τις αναγκαίες απλουστεύσεις και την ευελιξία για τα κράτη-μέλη και ότι αυτή η πρόταση διευκολύνει την επένδυση σε πολιτιστικές υποδομές και υποδομές για βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς να αμφισβητείται όλη η ισχύουσα, υπάρχουσα ε, ε, αρχιτεκτονική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά άλλους κανονισμούς που αφορούν την αξιολόγηση για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Νομίζω ότι το άλλο θέμα, το θέμα του τουρισμού και κατά πόσο ο πληθυσμός ζει από τον τουρισμό είναι ένα άλλο ζήτημα. Πρέπει να εξετάσουμε τις περιοχές όπου ο τουρισμός αναπτύσσεται τάσεις όσον αφορά τον τουρισμό, οι παρούσες τάσεις στον τουριστικό τομέα ε, δείχνουν και σημαίνουν ότι ο πληθυσμός ποτέ δεν θα μένει ανυπηρέαστος από το περιβάλλον. Ο η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του τουρισμού δεν θα πρέπει να εξαντλεί αλλά να συντηρεί τους πόρους για μελλοντικές γενναίες βελτιώνοντας συνθήκες διαβίωσης στον τόπο προορισμού. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μια πρόταση η οποία πρόταση θα πρέπει να δημιουργεί ε, σχέσεις μεταξύ του ΕΦΣΙ και του ΕΖΙΦ βάσει της προτάσεως ε, Omnibus και θα ήθελα η συγγήτρια να μας εξηγήσει ποια είναι η άποψή της, το όραμά της όσον αφορά τη συνύπαρξη των δύο ταμείων και τι συνέργειες μπορεί να υπάρξουν μεταξύ των δύο. Να κάνω κάποια σχόλια και εγώ για την έκθεση. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την κυρία Κρέλ γιατί η γνωμοδότηση αυτή έγινε υποπίεση. Υπό μεγάλη πίεση και χρονική και ε, προσδοκιών της ε, Καθήλυνα Ορμόδα Επιτροπής του Κοινοβουλίου. Οπότε έχουμε τώρα μια πρόταση γνωμοδότησης ε, της Επιτροπής Ρέτζη που είναι μια καλή βάση για συζήτηση και σίγουρα θα βρούμε από κοινού τις λύσεις. Καλωσορίζω φυσικά την πρόταση αυτή, γιατί αντικατοπτρίζει σε ένα μεγάλο βαθμό τι κοινέ προσπάθειε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Επιτροπή των Κρατών Μελών και, ενώ και όλων των εμπλεκομένων φορέων για την περαιτέρω απλούστευση τη ε, εφαρμογή των ε, διαφορετικών ταμείων και, ε, και το συνδυασμό με το ΕΦΣΙ και με τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα καθώς επίσης και της ε, μείωσης του διοικητικού άχθους προς τους επιλέξιμους. Επίσης, ε, ένα κομμάτι των τροποποιήσεων ε, αποτελεί αποτέλεσμα της δουλειάς που έγινε από την ομάδα υψηλού επίπεδου που δημιούργησε σχετικά η Κομισιόν. Αυτό έχει να κάνει με την απλούστευση. Εγώ ω σκιώδης θα ήθελα να υποστηρίξω τις τροπολογίε για τη μείωση του διοικητικού άκθους που σχετίζονται με τη χρήση των Ευρωπαϊκών Διορθωτικών Ταμείων επενδύσεων και επίσης συμφωνώ με την ε, εισηγήτρια για τις, ε, για τις ε, υποδομές μικρής κλίμακας που μπορούν να μείνουν στον κανονισμό για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης βάζοντας και ένα όριο ανώτατο. Αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις και γι' αυτό θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία για τον επαναπρογραμματισμό των προγραμμάτων και υποστηρίζω απολύτως την άποψή σας σχετικά. Υποστηρίζω επίσης τις προτινόμενες ε, τροποποίησεις του Omnibus ε, σχετικά με την απλούστευση των κανόνων και του συνδυασμού των ταμείων ΕΣΕΦ και των ε, χρηματοδοτικών μέσων για να υπάρξει συνέργεια και συμπληρωματικότητα που θα βοηθήσει την, ε, τον πλαπλασιασμό των επενδύσεων και θα κινητοποιήσει και την ιδιωτική χρηματοδότηση. Και επίση συμφωνώ και με τον κύριο Βανίστερόι που είπε ότι μέσω αυτών των συζητήσεων σίγουρα θα καταλήξουμε σε κάποια λύση. Γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε την ανάγκη που υπάρχει για νέε επενδύσει. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη διαδικασία της συμμετοχή των, των ιδιωτών επενδυτών. Οπότε πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα δύο αυτά μέσα. Ως προς αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε τις, πρωτο... τις προτάσεις ε, της που προτείνει η Κομισιόν χωρίς καθυστέρηση γιατί εάν αρχίσουμε να το αφήνουμε για τη μελλοντική, και περιμένουμε τη μελλοντική ε, νομοθετική πρόταση, θα περάσουν χρόνια συζητώντας. Ίσως να είναι λοιπόν καλό να χρησιμοποιήσουμε αυτή την επιλογή που έχουμε μέσω του Omnibus για να καταλήξουμε τελικά σε μια λύση για αυτό το θέμα της συμπληρωματικότητας. Αυτά είναι τα δικά μου σχόλια και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Βάνα που είναι η επόμενη σκιώδηση συγγετρία. Σας ευχαριστώ τα μάλα Κυρία Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω εκ βάθου στα καρδιά στην κυρία Κρέλ για την πρότασή τη, σύμφωνα σε πάρα πολλά σημεία τη γνωμοδότησή τη. Έχει παρουσιάσει μια γραμμή η οποία είναι πολύ θετική, ιδίω σε ό,τι αφορά την διαγραφή του άρθρου 30α που επιτρέπει την χωρίς περιορισμό μεταφορά κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία σε άλλες γραμμές του προϋπολογισμού. Έχω ήδη και σε άλλες ε, ευκαιρίες τονίσει γιατί κάτι τέτοιο αποτελεί μια πραγματική απειλή για την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απαραίτητο η Επιτροπή μας να πάρει μια σαφή θέση για το θέμα αυτό. Θέλουμε να υπάρξει και για το άρθρο 39α το CPR μια διαγραφή γιατί αυτό θα οδηγήσει σε μια επικράτηση των κανόνων του ΕΦΣΥ η οποία είναι πιο ασθενική. Είναι πιο αρνητική λοιπόν για αυτούς οι οποίοι επενδύουν. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα διατηρηθούν οι, φο... οι στόχοι της βιώσιμης πολιτικής και θα πρέπει να παραμείνουν αυτοί στο στόχαστρο Γι' αυτό το άρθρο 39α κινδυνεύει να επιδεινώσει την κατάσταση. Επίσης θα καταθέσουμε για κάποιες τροπολογίες για την ε, επιμερισμένη διαχείριση σε ό,τι αφορά τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό και την κοινή διαχείριση του ΕΣΥΦ με το ΕΦΣΥ, κάτι το οποίο το απορρίπτουμε εμείς θεωρούμε ότι η, η συνεργασία μεταξύ του ΈΣΥ και του ΕΦΣΥ δεν θα πρέπει να θίξει στο υψηλό επίπεδο της πολιτικής ε, συνοχής. Γι' αυτό έχουμε μία κριτική στάση σε ό,τι αφορά την ε, συνένωση αυτών των δύο εργαλείων πολιτικής. Εμείς βλέπουμε θετικά βέβαια και τις ε, αντιμετωπίσεις που αναφέρει η κυρία Κρέλ για την ε, αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ρεύματος και εγώ προσβλέπω σε μια ε, επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρτιν. Σας ευχαριστώ. Θα μπω στην ουσία του Omnibus και την πρόταση νομοθετική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όπως συμβαίνει και στην Ιταλία με τις διακηρύξεις, με τις παρατάσεις ε, ε, έχουν όλα σε ένα κείμενο, καλύπτονται τα πάντα. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε κάθε πτυχή της πρότασης από τις χορηγίες από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με τα δίκτυα της ευρωπαϊκά, τις υποδομές ψηφιακές ε, και τα παράσιτα των φυτών. Εδώ όμως ασχολούμεθα με αυτό που είναι αρμοδιότητά μας. Εκτιμώ το έργο της συναδέλφου Κρέλ και συμμερίζομαι πολλά από τα σημεία που τονίζει και συμφωνώ με την κατεύθυνση ε, που ακολουθεί και θα υποβάλω τροπολογίες. Το άρθρο 262 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει μια πιο ταχεία διαδικασία όσον αφορά την ένταξη της αλληλεγγύη στον προπολογισμό. Και είδαμε, όπως πρόσφατα, πόσο μεγαλύτερη ταχύτητα για τη διάθεση των πόρων μπορεί να είναι αποφασιστική σημασία για να βοηθούν οι πληθυσμοί που πλήττονται από φυσικέ καταστροφέ στα πλαίσια ενό μηχανισμού ε, συνέργειας μεταξύ εθνικών πόρων και ευρωπαϊκών. Στο άρθρο 264 προστίθεται στα πλαίσια του στόχου της προώθησης της κοινωνικής ένταξης η καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διακρίσεως η υποστήριξη της υποδοχής και της κοινωνικο-οικονομικής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων. Την άποψή μα όμω, η μετανάστευση δεν θα πρέπει να επιβαρύνει μοναδικέ περιοχέ και μοναδικά κράτη-μέλη. Συνεπώ, δεν θα έπρεπε να επιβαρύνει την πολιτική συνοχή. Το βάρο αυτή τη προβληματικής θα πρέπει να πέφτει στις πλάτες όλη τη Ένωσης με αποτελεσματικά κράτη και θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στην προσπάθεια. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με το 265 πέρα από το θέμα των εμπιστευμένων δαπανών και των χρηματοδοτήσεων κατά αποκοπή για το έμεσο κόστος για επιδοτήσεις και επιστροφή ενισχύσεων, ε, Όμω αυτό συνδυάζεται με κάτι που δεν μα αρέσει. Ενθιασμό του ΣΥΕΦ με το ΕΦΣΥ Δεν μα αρέσει αυτό. Ε, με προώθηση χρηματοσυντικών εργαλείων υψηλού κινδύνου και ε, προωθείται μια συνέργεια που αποκαλείται. Εγώ πιστεύω ότι το, το χρήμα που αφαιρεί την πολιτική συνοχή, ενώ οι πολιτικέ δομέ που κατασκευάζονται για την πολιτική κοινωνική και οικονομική και εδαφική συνοχή, αυτά τα έργα διαλύονται ή εξα, εξανεμίζονται ε, μέσα στη θολούρα του ΕΦΣΥ. Ε, θα πρέπει να δεχτούμε ότι το τμήμα που αφορά τεχνωστατικά εργαλεία, κυρίω ο συνδυασμό του ΕΦΣΥ με το ΣΥΕ, θα πρέπει να απορριφθεί. Διότι ουσιαστικά αυτό αντιστοιχεί σε απαράδεκτη αποδυνάμωση ε, τεράστια αποδυνάμωση της πολιτικής συνοχής, αν γίνει αυτός ο συνδυασμός. Thank Ευχαριστούμε πολύ. Άλλα σχόλια υπάρχουν? Όχι. Να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. And, the shadow rapporteurs. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την ε, εισηγήτρια την κυρία Κρέλ. Καταρχάς να ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνατε μέσα σε ένα τόσο σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Ο κοινό μας στόχος είναι να υιοθετηθεί η πρόταση όμνιμπος το συντομότερο δυνατόν όπως ξέρουμε όλοι. Συνολικά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ε, δουλειά που έχει γίνει και με το σχέδιο γνωμοδότησης. Βεβαίως ε, λυπούμε για την πρόταση που γίνεται να μείνουν εκτός όλα τα ανώτατα όρια ΕΦΣΙ και ΕΣΥΦ. Εμείς επιμένουμε να παραμείνουν οι διατάξεις αυτές εντός της πρότασης για να διευκολύνουμε την, το συνδυασμό των δύο έτσι ώστε να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο για το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν να γίνονται επενδύσεις και να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι από τη δική μας την οπτική είναι μια κατάσταση που βοηθά, ωφελεί και τους δύο και τα δύο ταμεία. Καταρχά, θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την ε, πρόσβαση των κονδυλίων, οπότε θα μπορέσουμε να έχουμε πιο ευνοϊκή ε, γεωγραφική κατανομή, ε, χρησιμοποιώντα ε, τα διαθετικά ταμεία για να μειώσουμε τον, το προφίλ κινδύνου κάποιων project, έτσι ώστε να μπορούν να προσελκύσουμε επιπλέον επενδύσει και να είναι πιο προσοδοφόρα τα διάφορα project για τις αδειγικές ας πούμε, επενδύσεις και το σχετικό ταμείο, αλλά και για τα διαρθρωτικά ταμεία, θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθήσει τις περιφερειακές αρχές, γιατί θα είναι σε θέση να έχουν περισσότερη δυνατότητα μόχλευσης ώστε να προσελκύσουν περισσότερες επενδύσεις ιδιωτικών φορέων για να καλυφθούν οι ανάγκες. Η διαθεσιμότητα λοιπόν των διαθετικών ταμείων κάποιε φορέ είναι πολύ περιορισμένη για να καλύψουν τα πάντα. Βεβαίω υπάρχουν πάντα ανάγκε εξήγηση και η Κομισιόν ευχαρίστω πάντα θέλει να έχει καλύτερη επικοινωνία μαζί σας για να δίνει τις διευκρινήσεις που χρειάζεστε. Κατανοώ ότι σε δύο ημέρες θα υπάρξει μια τεχνική συνεδρίαση με τα μέλη της Επιτροπής για να σας εξηγήσουμε με ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες ε, τον, ε, τα ωφέλη αυτού του συνδυασμού. Οπότε ελπίζω ότι αυτό θα είναι το πρώτο βήμα και βεβαίως είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για επιπλέον σχόλια και πληροφορίες. Το δεύτερο μου σχόλιο έχει να κάνει με το εξή. Με τη χρήση των ε, επιλογών για τα απλουστευμένα κόστη. Γιατί νομίζω ότι το συζητάτε στην Επιτροπή σα. Αυτό το θέμα είναι πραγματικά ένα θέμα που μα ενδιαφέρει ιδιαίτερω να υπάρξει δηλαδή η επιλογή υποχρεωτική ουσιαστικά τη χρήση των του απλουστευμένου κόστους γιατί θεωρούμε ότι αυτό υπό κάποιες προποθέσει μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απλούστευση του διοικητικού και μείωση του διοικητικού άκθου και για τις διαχειριστικέ αρχές. Βεβαίως εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας αλλά και πάλι λέω ότι όχι μόνο για την τρέχουσα πραγματική περίοδο, αλλά και για το μέλλον, είναι σημαντικό να προωθήσουμε αυτή την επιλογή, έτσι ώστε να πάμε σε μια κατεύθυνση που θα μας οδηγήσει τελικά σε μειωμένο διοικητικό βάρος για τις δραστηριότητε αυτές. Ε, σταματώ εδώ. Αν υπάρχουν ερωτήματα, ευχαρίστω να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος. Για να διευκρινιστεί για μένα. Μήπως μπορώ να σας ρωτήσω, αναφερθήκατε στην τεχνική, τεχνικού χαρακτήρα συνάντηση για την, ναι, ναι για την συγκεκριμένη. Ναι, κατάλαβα. Κυρία Κρέλα, έχετε τον λόγο. Και εγώ θα ήθελα πάλι να έχω κάποια βοήθεια από την Κομισιόν για να περιλάβω αυτά τα στοιχεία για, την, ε, για τις τροπολογίες. Πρέπει να γίνουν αυτές οι τεχνικές συζητήσεις που θα γίνουν, ε, η τεχνική συνάντηση που θα γίνει μεθαύριο για όλους τους ε, σκιώδεις εισηγητές για το θέμα αυτό, για την τεχνική πληροφόρηση από την Κομισιόν. Και υπάρχει δυνατότητα για διευκρινιστικές ερωτήσεις. Τώρα, Θέλω να σας αναφέρω ότι δεν θα ήθελα να παρακάμψουμε και να παραπέψουμε σε ελληνικές καλέντες το θέμα της σύνδεσης του ΕΣΥΦ και της ΕΦΣΥ Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο βέβαια να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα σε επίπεδο ουσίας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα στη διαδικασία του Omnibus. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι χώρε οι οποίες δίδουν ε, χρήματα για, την, ε, για τα ταμεία αυτά στην Κομισιόν θα έχουν την δυνατότητα να αποκομίσουν ωφέλη από τα χρήματα αυτά και επίση τα κράτη-μέλη αυτά θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι περιφέρειε οι οποίε θα ευεργετηθούν από αυτά τα σχέδια θα πρέπει να έχουν και κάποιο λόγο, κάποιο λόγο στη διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρό θέμα με πιο πολύ προσοχή από ό,τι μας δίνει η διαδικασία του όμιμπους. Δεν θέλουμε να το περάσουμε στα γρήγορα μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα πρέπει λοιπόν, δεν θα κάνω καμία τροπολογία για τα θέματα αυτά γιατί, που έχουν να κάνουν με την, ε, τις γραμμές του προϋπολογισμού. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο αφορά την Επιτροπή Προϋπολογισμού και Ελέγχου του Προϋπολογισμού και δεν μπορώ να τους κατηγορήσω για έλλειψη σοφροσύνης στα θέματα αυτά. Θα περιοριστώ στα θέματα που έχουν να κάνουν με την δική μας αρμοδιότητα ως Επιτροπής Περιφερειακών Θεμάτων. Δεν θέλω λοιπόν να εμποδίσω να προχωρήσουμε στην απλούστευση το ταχύτερο δυνατό. Επομένως, το θέμα της ε, ενσωμάτωσης του ΕΣΥΦ και του ΕΦΣΥ δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να εμποδιστεί, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη επίγνωση των προβλημάτων που συνδέονται με αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με προσοχή και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετό χρόνο στις 8 εβδομάδες που μας ε, ε, παραμένουν για την έγκριση του Omnibus να αντιμετωπίσουμε τα θέματα γιατί πρόκειται για πολλά χρήματα, πρόκειται για πολλές ε, επενδύσεις. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματικά εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και το θέμα αυτό με τους ε, Εγώ θεωρώ ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να βγει από τη διαδικασία που έχει να κάνει με το Omnibus. Θα πρέπει να εστιάσουμε πρώτα στο Omnibus και είναι απαραίτητο να έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε μεταξύ μας για το θέμα αυτό. Δεν πρόκειται για φιστίκια, δεν πρόκειται για ίσονα θέματα, θα πρόκειται για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και επέχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη και δεν μπορούμε να το περάσουμε ελαφρά την καρδία. Περιμένω λοιπόν από την Κομισιόν να μας δώσει και τις επόμενες μέρες και κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις για τα θέματα αυτά, γιατί καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι θέλουμε ότι έχουμε φτιάξει ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από ότι εξυπηρετεί την περιφερειακή πολιτική. Μπορεί η Κομισιόν να με μεταπίσει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε στον εαυτό μας τον χρόνο για να συζητήσουμε πλήρως και περισσότερο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Please, Mr. Προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη στη σχέση με το ΕΦΣΙ. Είναι σημαντικό, αλλά είναι και αναγκαίο να είναι ταχεία διαδικασία, γιατί όπως είπατε, πόσες φορές άκουσα από πλευράς Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να λέει ότι η ανάμιξη, το blending μπορεί να ισχύσει. Αυτή η ανάμιξη δύο διαφορετικών συστημάτων είναι κάτι ανόητο, απόλυτα ανόητο, διότι δημιουργούνται πολλά προβλήματα για τους δικαιούχους αργότερα έχει το ένα ή το άλλο σύστημα. Αντί να είμαστε ακριβέστεροι, δεν είμαστε. Ίσως σε αυτή την νομοθεσία να δείχνουμε κάποιες κατευθύνσεις και μετά έχουμε παράταση του έψι Ξεχωριστή διαδικασία. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι να κάνουμε κάτι σε ένα βήμα και κάτι να επιστρέφει. Δεν είναι ανάμιξη. Παίρνουμε χρήματα από τα ταμεία συνοχής και τα βάζουμε σε άλλο εργαλείο, στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ. Ποιες εγγυήσεις έχουμε ότι θα επιστρέψουν στις περιφέρειες τα χρήματα. Αυτά τα πράγματα είναι προβληματικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μετά το 2020. Πρέπει να το προθήσουμε. Αν παρόμοια με το ΕΦΣΥ εργαλεία συνεχιστούν οι χώρες μπορεί να πούν επιλέγουμε μία εύση μεθοδολογία και μπορεί να είναι σημαντικό για μία χώρα και όχι για άλλη. Πώς να το πω, την υπόλοιπη περίοδο τη χρησιμοποιούμε για να δούμε τι γίνεται με ένα σύστημα. Αν δεν μπορούμε να καθορίσουμε τι θέλουμε, ποιος μπορεί να το καθορίσει. Μπορούμε να υπερασπιστούμε την προσέγγιση του Ταμείου Συνοχής, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ και πιθανότατα στην παράταση του ΕΦΣΙ θα πρέπει να καθορίσουμε αυτή την εδαφική προσέγγιση. Διότι τώρα στην αξιολόγηση Όσον αφορά το ΕΦΣΙ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ναι, ναι, πρέπει να βρούμε καλύτερη εδαφική ισορροπία. Ίσως μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Ας καταφέρουμε να βγάλουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε τώρα βραχυπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι η αυριανή συνεδρία θα είναι άκρο ενδιαφέρουσα και καρποφόρα. Συνεχίζουμε αύριο αυτή τη συζήτηση. Έχουμε τη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών αύριο. Και εκεί μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, ευχαριστώ για την πρόταση. Να επενθυμίσω ότι έχουμε 7 μέρες για την εκνοή της προθεσμίας υποβολής τροπολογιών. Επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως, τα διάφορα. Δεν υπάρχουν διάφορα. Να σας υπενθυμίσω, η επόμενη συνεδρίαση, Δευτέρα, 20 Μαρτίου, από τις 3 το απόγευμα, ξεκινάμε, και την Τρίτη, 21 Μαρτίου, από τις 9 την πρωιέν. Και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 18.30 το απόγευμα πέρας του δημοσίου τμήματος των συζητήσεων της Επιτροπής μας και θα συνεχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε, αυτοί που δεν δικαιούνται να παρίστανται συνεδρίαση των συντονιστών παρακαλώ να αποχωρήσουν από την αίθουσα.